je vous propose de commencer euh, nos travaux puisque nous devons recevoir euh, la présidence espagnole euh, dans quelques dizaines. Ας αρχίσουμε με Είχαμε μια μικρή καθυστέρηση. Είχαμε βέβαια τα πορίσματα της συνάντησης των συλλογιστών από χθες. Καταρχήν η κυρία Ντεβεράκ μας μίλησε για την συμφωνία στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Όλα τα σημεία στα οποία πέτυχε συμφωνία τα δέχονται οι συντονιστές και θα ψηφιστούν στις 2 Σεπτεμβρίου από την Επιτροπή μας. Η ψηφοφορία της έκθεσης για τα ατυχήματα και διάφορα επεισόδια που συμβαίνουν σχετικά με την αεροπορία προβλέπεται για τις 11 Συγγνώμη. 2 Σεπτεμβρίου. 10 Σεπτεμβρίου μάλλον λέει ο πρόεδρο. Επίσης συζητήσαμε για τον ορισμό εισηγητών. Πρώτη έκθεση. Η Ευρώπη ως πρώτος τουριστικός προορισμός. Νέα πολιτική ατζέντα για τον τουρισμό στην Ευρώπη. Ομάδα του ΕΛΚΑ. έκθεση γνωμοδότησης για μια σύνθεση σχετικά με τα πορίσματα του management της Κομισιόν για το 2009 δεν θα γίνει έκθεση. Έκθεση της Επιτροπής Κομισιόν για την Πολιτική Ανταγωνισμού 2009. Η απόφαση είναι η ομάδα που θα την πάρει θα είναι το ΕΛΚ. Τελικά όμως έγινε μια ανταλλαγή μεταξύ των Πρασίνων και του ΕΛΚ. Οι Πράσινοι θα πάρουν την έκθεση για τον ανταγωνισμό, πολιτική ανταγωνισμό του 2009 σε αντάλλαγμα με μια ανακοίνωση για τη στρατηγική για τα καθαρά και αποδοτικά σε ενέργεια οχήματα που ήταν έκθεση των Πρασίνων αρχικά. έκθεση για ένα πρόγραμμα δράσης για τα συστήματα πλοηγισμένου αδερφόρου NSS με ιδιαίτερη εστίαση σε θέματα μεταφορών αλληλιστές δημοκράτες. Έκθεση για την εφαρμογή πολιτικής συνοχής πρόγραμμα του 2007 2007-2013, ήταν η προσωρινή έκθεση, η Γνωμοδότηση είναι αυτή. Και τέλος, η ομάδα EFD ε πήρε την έκθεση για την European Agenda Έβδομη έκθεση πρωτοβουλίας για τις διεθνείς ε, συμφωνίες για τα αεροπορικά με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτό θα τον κάνει ο πρόεδρος καμία ομάδα δεν επέδειξε ενδιαφέρον. Ο πρόεδρος πληροφόρησε τους συντονιστές για την αύξηση των δαπανών για τους συντονιστές για τα FABs και ορίστε ο κύριος Γιαρζεμπόφσκι ως συντονιστής για τα θέματα τα αεροπορικά. Επίσης αναφέρθηκε η άλλη πληροφορία ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια διαφορά μεταξύ Ουκρανίας και της Austrian Airlines που κατά κάποιο τρόπο τις αφαιρέθηκαν μονόπλευρα τα σλότ που είχε στο αεροδρόμιο του Δνίπε Πετρόφσκ αλλά γίνονται διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή δεν το κατάλαβα ακριβώ πόσο τόσο κάτι τέτοιο συμβαίνει. Το θέμα για τα κοντέινερ που χάνονται στη θάλασσα Βαντέλεν θα αποτελέσει αντικείμενο προφορικής ερώτησης που θα τεθεί από την Κομισιόν εκτός να το κάνει ο Αντιπρόεδρος. Προφορική ερώτηση για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες που ήταν αντικείμενο και πρόταση του Πρόεδρου και συζήτηση από τις ομάδες θα τεθεί ως έχει διότι οι συντονιστές δέχτηκαν το κείμενο ως έχει μετά είχαμε ανταλλαγή απόψεων, αναφέρθηκε και αυτό. Ε, συγγνώμη, ανταλλαγή επιστολών. Ιδιαίτερα μια επιστολή σε δρυμή ύφο. σε έντονο ύφο που ειστάγει από τον πρόεδρό μα. για την αναθεώρηση του πρώτου σιδηροδρομικού πακέτου σε σχέση πάντα με την παρέμβαση μιας χώρας ως προς τον, την Κομισιόν, προς τον πρόεδρο της Κομισιόν μάλιστα και μια διαμαρτυρία που την προσυπέγραψαν όλοι οι συντονιστές γιατί είναι απαράδεκτο μια μεταφορά αυτής της αναθεώρησης του σιδηροδρομικού πακέτου να γίνει ιδιαίτερα κάτω από αυτές τις συνθήκες. Επίσης πήρε μια επιστολή της κυρίας Ντιρόν για τη συνεδρίαση των πολιτών για το Αγκορόκ, για την φτώχεια και ζητούν συμβολή της Επιτροπής μας. Η κυρία Ντυρό θα έρθει στην συνεδρίασή μας στις 2 Σεπτεμβρίου να μας εξηγήσει τι ακριβώς περιμένουν από μας. Επίσης είχαμε πληροφόρηση για την ομάδα ΣΤΟΑ και την πρόταση για τις προθεσμίες για τις συμβαστικές τροπολογίες. Θα υπάρχουν δύο είδη εκθέσεων πέραν τροπολογιών, πολλές τροπολογίες, πάνω από 50 τροπολογίες θα θεωρείται ότι χρειάζονται επιπλέον τρεις εβδομάδες πριν ψηφιστεί στην Επιτροπή προκειμένου να επιτευχθούν συμβιβασμοί για να μειωθούν οι τροπολογίες. Στην αντίθετη περίπτωση θα ισχύσει η συνήθις διαδικασία. Συζήτηση στην Επιτροπή και ψηφοφορία την επομένη. Ο κύριος Κράμερ ανάφερε ένα πρόβλημα με τις γραμμές των τρένων στην Ελλάδα που έκλεισαν ενώ είχαν χρηματοδοτηθεί με κοινωτικά κονδύλια, ευρωπαϊκά κονδύλια. Είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα αυτό. Πρέπει να τεθεί. Συμφωνήθηκε να υπάρξει μια παρέμβαση στην Κομισιόν για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Ο κ. Σαλκαντράουι ζήτησε και το κάλυψε και ο πρόεδρος το θέμα αυτό για να συζητηθεί η επόμενη επίσκεψη της αντιπροσωπείας για τον επόμενο χρόνο από 5 σε 3 και ενδεχομένω να αυξηθούν οι συμμετέχοντες μέχρι τότε ήταν περιορισμένο σε 5 να έχουμε περισσότερες επισκέψεις μάλλον λιγότερες επισκέψεις και περισσότερους συμμετέχοντες. Εν πάση περιπτώσει αυτό θα το ξανασυζητήσουμε όπως επίσης και η οδηγία για το ε, Ευρωβινιέτ. Ο κύριος Γκρός, και αυτό θα το συζητήσουμε σίγουρα πολύ, πρότεινε να συζητηθούν το θέμα των περιφερειακών ταμείων συνοχής και διορθωτικά δηλαδή και το πώς εφαρμόζονται στις επενδύσεις για υποδομή μεταφορών να προτείνουμε κοινή επιτροπή προκειμένου να προλάβουμε ορισμένες εντάσεις ορισμένες διαφωνίες, παραφωνίες που μπορεί να σημειωθούν για ένα θέμα που αποτέλεσε αντικείμενο τροπολογίας της έκθεσης του κ. Ρώσ για το μέλλον των μεταφορών που στη δική μας Επιτροπή είχαμε κοινή συμφωνία το θέμα αυτό δηλαδή παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για πολλούς και θα μπορούσαμε να το δούμε από κοινό όπως σας είπαμε Επιτροπή με την Επιτροπή Περιφερειών. Αυτά είχα να πω, δεν ξέρω αν θέλετε εξηγήσεις σχόλια, Μάικελ. Δεν ξέρω αν υπήρξε κάποιο πρόβλημα με την ε, μετάφραση μόλις τώρα. Δεν είπαμε ότι προφορική ερώτηση θα θέσουμε. Διακόπτει ο κύριος σκάμε. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν υπήρξε κάποιο πρόβλημα με τη μετάφραση, ε, αλλά σε ό,τι αφορά το ζήτημα της Ελλάδας είπαμε πως ε, γραπτή επερώτηση θα θέσουμε, όχι προφορικά. Ε, απλά σα λέω το άκουσα από αυτό από τη διερμηνία και ήθελα να το διευκρινίσω. Ο κύριο Σίμψον λοιπόν γραπτό θα απευθυνθεί σε σχέση με αυτό. Ναι, ναι, αυτό είπα και εγώ. Να γράψουμε επιστολή προ την Κομισιόν και να ζητήσουμε πληροφορίε. Όχι προφορική ερώτηση, επιστολή προ την Κομισιόν. Γιατί χρειαζόμαστε πληροφορίε για μια συγκεκριμένη χώρα. Δύο συνδρομικέ γραμμέ περί αυτού πρόκειται. Άλλε ερωτήσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια διευκρίνηση. Αναφερθήκατε στη δυνατότητα συγχρηματοδότησης προγραμμάτων ε, μεταφορών για τα διευθυντικά ταμεία και τομείες συνοχής. Μπορεί να πείτε κάτι παραπάνω. Τι λέει η πρόταση συγκεκριμένα. Γιατί εγώ είμαι και στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και με ενδιαφέρει το θέμα, αλλά δεν κατάλαβα καλά. Τι λέει η πρόταση. Πρόεδρος. Είπα με πολύ πολύ προσοχή προσεκτικό στα λόγια μου προτάθηκε και ελπίζω να γίνει δεκτό σε μέλη της ε, Περιφερειακής Επιτροπής να συναντηθούν με την Επιτροπή Μεταφορών για να συζητήσουμε τα της εφαρμογής και ζηγίζω τα λόγια μου την εφαρμογή των περιφερειακών ταμείων στην χρηματοδότηση των ε, δικτύων που έχουν προτεραιότητα RTET. Μόνο για την εφαρμογή τους, γιατί, de facto ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι περίπου 20 δις ευρώ των περιφερειακών ταμείων χρησιμοποιούνται για το RTET. Το να συζητήσουμε το αν θα μπορούσε ενδεχομένω να αφαιρεθούν ε, κυριαρχικά δικαιώματα οι ευθύνε από την Επιτροπή Περιφερειών Διαχείρισης των Κονδυλίων. Να δούμε ταυτόχρονα πώς μπορούμε να συμφωνήσουμε με την Επιτροπή Περιφερειών προκειμένου να πετύχουμε την optimum χρήση αυτών των κονδυλίων. Ξέρω ότι η Περιφερειακή Επιτροπή ανησυχεί για το εξή ότι να γίνει ένα είδος κατάσχεση ενός τμήματος των κονδυλίων αυτών προς ένα ταμείο για τις μεταφορές. Δεν Πρόκειται περί αυτού. Το θέμα είναι πώς θα μεγιστοποιηθεί η δράση των κοινωνικών κονδυλίων. Έχετε το λόγο, συνάδελφε. Για να δω αν κατάλαβα. Μήπως υπάρχει πρόβλημα μετάφρασης. Εγώ αυτό που άκουσα είναι το εξή. Αναφέρεται στην Επιτροπή Περιφερειών, όχι στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αυτό άκουσα από τα αγγλικά. Αναφέρεστε στην Επιτροπή Πολιτικής Περιφερειακής Ανάπτυξης Πρόεδρος. Αναφέρθηκα στην Επιτροπή, την Περιφερειακή Επιτροπή. Όχι την Επιτροπή των Περιφερειών. Όχι στην Επιτροπή των Περιφερειών. Άλλες ερωτήσεις ή σχόλια. θα πρέπει να περιμένουμε την Ισπανική Προεδρία όπου να ανέρχεται στις 9.30 μάλλον να μας κάνει τον απολογισμό της Ισπανικής Προεδρίας για τις μεταφορές και το αντίστοιχο συμβούλιο και το απόγευμα θα έχουμε τη Βελγική Προεδρία και τον ε, Υφυπουργό Μεταφορών και την Υπουργό Τουρισμού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 Κυρίες και κύριοι, έχουμε την ευχαρίστηση να υποδεχτούμε τον κύριο Μπλάνκο, ο οποίος είναι υπουργό Μεταφορών της Ισπανίας, ε, είναι και υπουργό και των πρωταθλητών, των παγκοσμίων πρωταθλητών. Έτσι, να το τονίσουμε αυτό. Κύριε Υπουργέ, Ολοκληρώνετε την εξάμενη προεδρία σας. Σας ευχαριστούμε που παρευρίσκεστε εδώ για να μας παρουσιάσετε το αποτέλεσμα των εργασιών σας και να απαντήσετε στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια στην καλύτερη ομάδα του κόσμου. Πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ και πάλι να παρευρεθώ εδώ σήμερα, στον οίκο αυτό, για να σας ε, παρουσιάσω μια αποτίμηση των κύριων δράσεων που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου της ε, Ισπανικής Προεδρίας του Συμβουλίου Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως σας παρουσίασα την ε, πρώτη μου εμφάνιση εδώ τον Ιανουάριο, Κατά τη διάρκεια αυτού του εξωμήνου, η Ισπανική κυβέρνηση είχε θέσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα προτεραιοτήτων και ήδη σας παρουσιάζεται τα πρώτα αποτελέσματα τη δεύτερη φορά που παρουσιάστηκα εδώ σε αυτό τον οίκο στα τέλη Μαρτίου. Αξιότιμοι κύριοι, πιστεύω ότι με τη βοήθεια και τη συνεργασία της Κομισιόν, με τη βοήθεια και τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πετύχαμε τα, στους περισσότερους από τους στόχους που είχαμε θέσει. Επίσης, ε, η προώθηση ε, ορισμένων των στόχων αυτών ενισχύθηκε ως συνέπεια των ε, συμβάντων που έλαβαν χώρα τους τελευταίους μήνες. Όπως φαντάζεστε, αναφέρομαι στην πρωτοφανή κρίση που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε στο ευρωπαϊκό εναέριο χώρο ως συνέπεια της έκρηξης του Ισλανδικού Εφεστίου τον περασμένο Απρίλιο. Και εκεί επικεντρώσαμε τις προσπαθίες μας το δεύτερο σκέλος του εξαμήνου και για πρώτη φορά έκλεισαν οι Ευρωπαίοι ουρανοί από το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Κατά τη διάρκεια της κρίσης, η Ισπανική Προεδρία, σε συνεργασία με την Επιτροπή και με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, από πρώτη πρώτη στιγμή ενεργοποίησε όλους τους μηχανισμούς προβλέποντας τον Ευρωκοντρόλ, πάντοτε ως, ε, έχοντας ως προτεραιότητα διαπραγμάτευση την εγγύηση της ασφάλειας. Επίσης, καλέσαμε δύο έκτακτες συνεδριάσεις του Συμβουλίου Μεταφορών στις 19 Απριλίου μέσω τηλεδιάσκεψης και στις 4 Μαΐου. Οι συναντήσεις αυτές μας επέτρεψαν να απαντήσουμε συντονισμένα στην κρίση. Αφού επιλήθηκε η κατάσταση, θεωρήσαμε ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή να προβληματιστούμε για την απάντηση που δόθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην κρίση αυτή και γι' αυτό αποφασίσαμε να εκπονήσουμε μαζί με την Κομισιόν συμπεράσματα που εγκρίναμε στο Συμβούλιο των Υπουργών στις 24 Ιουνίου όπου περιλαμβάνονται διάφορα μέτρα για τη βελτίωση της διαχείρισης σε παρόμοιες κρίσεις. Μεταξύ αυτών είναι και όταν αναπτυχθεί μια νέα επιστημονική τεχνική επιστημονική μέθοδος για την αξιολόγηση των κινδύνων, για την ασφάλεια σε περιπτώσει κρίσεων είναι και θα να διασφαλίσουμε το μέγιστο τα δικαιώματα των επιβατών ε, εφαρμόζοντας την υφιστάμενη νομοθεσία και λαμβάνοντας υπόψη τα διδάγματα που προέκυψαν από την κρίση τη σημασία τη ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού σχεδίου κινητικότητας για να εφαρμόζεται από τα κράτη-μέλη σε περίπτωση που έχουμε παρόμοια κρίση και η σημασία να δίνουμε μέγιστη προτεραιότητα στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ουρανού με δράσεις όπως η δημιουργία ενός ε, συντονισμένου κέντρου κρίσεων ή το διορισμό ενός διαχειριστή του Ευρωπαϊκού Δικτύου πριν τα τέλη του 2010 ή την επιτάχυνση των ε, ε, της ανάληψης των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού τη ασφαλεία τη αερομεταφορά. Όπω ξέρετε, η πρόθεση τη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ενίου Ουρανού ήταν ένα από του κύριου στόχου τη Προεδρία μα, στι 26 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο τη συνδιάσκεψης που κάλεσε η Ισπανική Προεδρία και η Επιτροπή, εγκρίθηκε η αποκαλούμενη δήλωση της Μαδρίτης και εκπονήθηκε ο δικός χάρτης για να επιτεχύνουμε την οριστική εφαρμογή ενός πραγματικού ευρωπαϊκού ενιαίου ουρανού που όπως σας είπα θα επιτεχυνθεί ακόμη περισσότερο ως συνέπεια της κρίσης του ηφαιστείου. Με την πλήρη εφαρμογή του θα μειωθούν από 69 ο αριθμός των κέντρων ενέργειων ελέγχων στον ευρωπαϊκό χώρο ε, και η αυτό μαζί με τη χρήση του συστήματος ΣΕΣΑΡ θα μας επιτρέπει να μειώσουμε στο μισό το κόστος των ε, τιμών ε, των οδών των πτήσεων, να μειώσουμε κατά 10% τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο και να βελτιώσουμε την επίπεδο της ασφάλειας. Επίσης, θα υπάρξει μείωση του κόστους περίπου 5,5 δις για τις ευρωπαϊκές εταιρείε, για του ευρωπαϊκού αερομεταφορεί. Και αυτό σημαίνει ότι θα βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά του και αποδοτικότητά του. Κατά τη διάρκεια του περισμένου εξάμεινου, Αναφέρθηκα πολλές φορές στο ότι η Ευρώπη μπόρεσε να αποκτήσει ενιαία αγορά και ενιαίο νόμισμα, αλλά ακόμη δεν είχε ένα ενιαίο ουρανό. Τώρα βρισκόμαστε πολύ κοντά στην επίτευξη αυτού του στόχου. Πιστεύω ότι τελικά μετατρέψαμε μια μεγάλη κρίση σε μια ευκαιρία για να δώσουμε ένα, ε, μια μεγάλη όθηση στην ε, υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ουρανού. Επίσης, ε, έχω επαναλάβει ότι το να έχουμε ένα κατάλληλο ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών σήμερα είναι κάτι πιο προφανές παρά ποτέ. Μεταξύ των προτεραιοτήτων μας ε, υπήρξε η εγγύηση να έχουμε ένα σταθερό και διασυνδεδεμένο δίκτυο μεταφορών στην Ευρώπη, ε, η Ισπανική Προεδρία, σε συνεργασία με την Κομισιόν, οργάνωσε στις 48 8 και 9 Ιουνίου ε, μία συνεδρία με στόχο να αναλύσουμε το, μέλλον, το παρόν και το μέλλον των διευρωπαϊκών ε, δικτύων μεταφορών το έγγραφο που υιοθετήθηκε από την Κομισιόν στις 4 Μαΐου και οι Γενικές Αρχές ε, είναι κάτι το οποίο βρίσκουν απόλυτα σύμφωνα την Ισπανική κυβέρνηση. Θέλουμε να τονίσουμε την διατροπικότητα την ε, βελτιστοποίηση του κόστους και την περιβαλλοντική εφορία αφού θα έχει επικυρωθεί η μεθοδολογία και υπάρχει και κατάλληλη συνένεση μεταξύ των κρατών, θα αρχίσουμε να ε, χαράζουμε τους άξονες και τους διαδρόμους που θα συμπεριληφθούν στο μελλοντικό βασικό ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών. Έτσι, ε, λοιπόν, το ενδιαφέρον της Ισπανίας ε, στο μεσογειακό διάδρομο συμπεριλαμβάνεται αυτό το project ως ένας στρατηγικός κρίκος ε, για ε, τις υποδομές των μεταφορών. Επιπρόσθετα, προωθήσαμε ένα προβληματισμό για την αναγκαιότητα να μελετήσουμε την ε, δυνατότητα δημιουργίας νέων ταμείων ή να ενισχύσουμε τα υφιστάμενα. Έτσι λοιπόν θα ήταν καλό να αξιολογήσουμε τη βιωσιμότητα, οι πόροι που έχουν ε, χρησιμοποιηθεί για τα διευρωπαϊκά δίκτυα να μην θεωρηθούν ως δημόσιο έλλειμμα σε σχέση με την υλοποίηση των στόχων του προγράμματος σταθερότητας. Επίσης, κάναμε πολύ σημαντικά βήματα σε ό,τι αφορά την απελευθέρωση των υπηρεσιών και της διεθνούς συνεργασίας. Προ την κατεύθυνση αυτή, θεωρώ πολύ μεγάλη επιτεύξη την υπογραφή του δεύτερη φάση τη συμφωνία για τι ενέργειε μεταφορέ μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένων Πολιτειών, που έλαβε χώρα στις 24 ε, του, μη, του περισμένου μήνα στο Συμβούλιο του Λουξεμβούργου. Κατά τη διάρκεια αυτού του εξαμήνου υλοποιήθηκαν τρεις από τους οκτώ γύρους που χρειάζονται για την υλοποίηση της συμφωνίας ε, που ξεκίνησαν από το 2007. Οι συνεδρίες αυτές έγιναν υπό Ισπανική Προεδρία και θα ήθελα να τονίσω ε, τη συνεισφορά της Κομισιόν, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και του κυρίου Λαχούντ που είναι ο Αμερικανός Υπουργός Μεταφορών. Ε, η συμφωνία αυτή θα διευκολύνει ε, μεγαλύτερη προσέγγιση μεταξύ Ευρωπαίων και Αμερικανών πολιτών, θα διευκολύνει το διάνοιγμα νέων οδών με καλύτερες και περισσότερες προσφορές και θα επιτρέψει τη δημιουργία περισσότερων θέσεων απασχόλησης και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και οικονομική μεγέθυνση. Επίσης, στις 18 Ιουνίου ε, και ένα μνημόνιο ε, συνεργασίας σε ό,τι αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη με την Ομοσπονδιακή ε, Υπηρεσία Αερομεταφορών των ΗΠΑ. Ως ε, κύριο στόχο έχει το ΣΕΣΑΡ να είναι συμβατό με το Αμερικανικό πρόγραμμα Next Gen. Επίσης, η πρόθεση της πολιτικής απελευθέρωσης και συνεργασίας μας επέτρεψε στις 24 ε, του Μαΐου να υπογράψουμε στο Rio de Janeiro μια κοινή δήλωση μεταξύ Βραζιλίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί καταγράφουμε την πρόθεση και των δύο μερών να υπογραφεί μια οριζόντια συμφωνία για τις ενέργειες υπηρεσίες και μια συμφωνία για την επιχειρησιακή ασφάλεια. Η υπογραφή αυτή θα λάβει χώρα πιθανότητα στη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Βραζιλίας που θα λάβει χώρα αύριο. Είμαι σίγουρος ότι αυτή η ορμή θα μεταφραστεί σε μια συμφωνία επίσης με τη Βραζιλία για τον ανοιχτό ουρανό. Επίσης, ε, κάτι άλλο που, πέτυχε η Προεδρία μας ήταν η πρόθεση ενός συνόλου μέτρων σε ό,τι αφορά την ασφάλεια. Έτσι λοιπόν, σε πρώτη ανάγνωση καταλήξαμε στη συμφωνία μαζί σας για τον κανονισμό, για την έρευνα και την πρόληψη των ατυχημάτων στην ε, πολιτική αεροπορία που θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα να τονίσω ότι εισαγάγει την υποχρέωση διαβίβασης καταλόγων επιβατών στις αρμόδιες αρχές μετά από κάποιο ατύχημα μέσα σε 12 ώρες. Έτσι αποφεύγουμε ε, τις ε, καθυστερήσεις που προκύπτουν μετά από ένα ατύχημα. Επίσης, η Κομισιόν παρουσίασε μία έκθεση για τα σκάνερα ασφαλείας, την συνέπειές του στην υγεία και άλλα θεμελιώδη δικαιώματα όπως και τον οικονομικό αντίκτυπο. Κατά την τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου Μεταφορών συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε να μελετάμε τα διάφορα μέτρα που προτείνονται από την Κομισιόν έτσι ε, ώστε στην περίπτωση υλοποίησης να έχουμε ε, ένα αρμονισμένο, μια εναρμονισμένη εφαρμογή έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουμε και τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν στους χρήστες στη συνεδρίαση στην Ακορούνια ε, συζητήσαμε μία αστική βιώσιμη και αποτελεσματική κινητικότητα μέσω της προώθησης ε, των ε, δημοσίων μεταφορών. Εγκρίναμε ομόφωνα στις 24 Ιουνίου συμπεράσματα του Συμβουλίου για την αναγκαιότητα να συντονίσουμε τη δράση των δημοσίων διοικήσεων σε κοινοτικό περιφερειακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο για να διευκολύνουμε την εφαρμογή σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητα και να προωθήσουμε τις δημόσιες μεταφορές και Επίσης, η Ισπανική Προεδρία προώθησε μεταξύ άλλων τις εργασίες για να εγκρίνει τον κανονισμό για τα δικαιώματα των επιβατών που ταξιδεύουν με λεωφορεία. Και ελπίζουμε ότι για το κείμενο αυτό, πέρα από τα εκρεμή ζητήματα, θα καταλήξουμε σε οριστική συμφωνία σύντομα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, κάναμε μια σημαντική προσπάθεια στη διαπραγμάτευση του κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών που ταξιδεύουν ε, στη θάλασσα και δια των πλωτών εδών. Και αυτό μας επέτρεπε να καταλήξουμε συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση που κυρώθηκε ε, στις 6 του μήνα στην Ολομέλεια από το Κοινοβούλιο και αυτό θα σημαίνει ότι θα έχουμε σημαντική πρόοδο κυρίως για τα άτομα με ειδικέ ανάγκες και με περιορισμένη κινητικότητα. Τώρα θα σας ενημερώσω για άλλου ε, φακέλους ε, με τους οποίους ασχολήθηκε η Προεδρία μας. Η Προεδρία έκανε το απαραίτητο έργο για να εγκρίνει τον κανονισμό για το σειροδρομικό δίκτυο, για τη μεταφορά ε, των αγαθών. όπω ξέρετε, Συμβούλιο και Κοινοβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία. Έτσι λοιπόν τώρα το Συμβούλιο κατά τη διάρκεια τη Βελγική Προεδρία πρέπει να εγκρίνει το συμφωνημένο κείμενο. Σε ό,τι αφορά τώρα ε, τη θαλάσσια ασφάλεια, καταλήξαμε σε μια συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση για την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις απαιτούμενες διατυπώσεις από τα σκάφη όταν ε, ε, καταφθάνουν ή αναχωρούν απολυμμένες. Επίσης, καταλήξαμε σε μια συμφωνία για την ε, οδηγία για το φορητό εξοπλισμό πίεσης. Η οδηγία αυτή δημοσιεύτηκε στις 30 Ιουνίου στην επίσημη εφημερίδα. Τώρα, να αναλύσω άλλου από του κύριου στόχου που προώθησε η δική μα Προεδρία. Θα ήθελα να σα ενημερώσω για την πρόοδο στην καινοτομία. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα Γαλιλαίο, υλοποιήσαμε μια συμφωνία, συνάψαμε μια συμφωνία συνεργασία για την Νορβηγία και δώσαμε εντολή στην Κομισιόν για να ξεκινήσει τι διαπραγματεύσει με την Ελβετία. Και σε αυτό το δεύτερο εξάμεινο προβλέπεται και άλλε δράσει, όπω ενδιάμεση αναθεώρηση του προγράμματο. Επίση, πρέπει να τονίσουμε ότι καταλήξαμε καταλήξαμε σε μια συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση για την τροποποίηση του κανονισμού 1321-2004 του Συμβουλίου σε σχέση με τις δομές διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ραδιοπλοήγησης μέσω δορυφόρου και σε σχέση με τα έξυπνα συστήματα μεταφορών, πρόταση οδηγία ε, για τη δημιουργία ενός πλαισίου για την εγκατάσταση των συστημάτων, ε, έξυπνων συστημάτων μεταφορέ για τις μεταφορές. Εκεί καταλήξαμε σε μία πρώιμη συμφωνία, στη δεύτερη ανάγνωση, που επίσης εγκρίθηκε στη τελευταία ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 6 του μήνα. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ολοκληρώσω τώρα την παρέμβασή μου τονίζοντας ε, το ότι είχαμε εξαιρετική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Κάλλας, καθώς και με τις υπηρεσίες της Κομισιόν συνεργασία αυτή ήταν ε, επίσης πολύ εντατική με τους υπόλοιπους ε, ομολόγους μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ε, επίσης και με τα μέλη αυτής της Επιτροπής και με τον Πρόεδρο, τον κύριο Σίμψον, ο οποίος απουσιάζει σήμερα. Όλες τις δράσεις αυτές που αναπτύξαμε στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων που καθορίστηκαν από το τρίο των Προεδριών, είμαι σίγουρος ότι θα συνεχιστούν από τη Βελγική και την Ουγγρική Προεδρία. Θα ήθελα να τους ευχηθώ κάθε επιτυχία τις εργασίες τους και γιατί αν είναι επιτυχής οι προεδρίες αυτές θα αποτελέσει και αυτό επιτυχία για το σύνολο της Ένωσης υλοποιήσαμε μια φιλόδοξη ε, ατζέντα με πολύ σημαντικά θέματα για τη βελτίωση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφορών και γι' αυτό πιστεύω ότι τα αποτελέσματα που, αποκτήθηκαν με συγχωρείτε στο εξάμεινο αυτό αποτελούν πρόοδο για την επίτευξη μιας πιο ολοκληρωμένης και αϊφόρου πολιτική μεταφορός που θα εξυπηρετεί τους Ευρωπαίους πολίτες. Σας ευχαριστώ. Euh, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ για την ενδελεχή αυτή παρουσίαση του απολογισμού της Προεδρίας σας. Το λόγο στους συντονιστές των ομάδων με τυχόν ερωτήσεις ή σχόλια. Κόντες Πασκάλ, ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλωσορίσατε στον οίκο αυτό. Νομίζω ότι είναι η τρίτη φορά που έρχεστε εδώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω λοιπόν για τη στάση που έχετε απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κύριε Υπουργέ, Όταν ε, εσείς ε, παρουσιάζεστε ως ε, τεχνοκράτης, ξέρετε, εγώ το κατανοώ, αλλά μπορώ να σας πω ότι μάλλον λαμβάνετε διαφορετικό ρόλο το Σαββατοκύριακο όταν παίζατε με τους Ολλανδούς. Κοιτάξτε, εγώ τώρα να σας πω ότι εδώ θα είμαι ευγενικός μαζί σας γιατί έχουμε κερδίσει και το πρωτάθλημα, το κύπελο. Θα ήθελα να σας πω ότι ήταν αποτελεσματικό το έργο σας ε, και να σας πω ότι η Ισπανική ομάδα ε, είναι εξαιρετική και αναφέρομαι στη μόνιμη αντιπροσωπεία. Έχουμε και τον συνάδελφο που κάθεται δίπλα σας, θα πρέπει να τον ευχαριστήσουμε. Πραγματικά πρέπει να σας ε, αναγνωρίσω το έργο σας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια χώρα. Είστε πολύ συνεπείς. Αναφερθήκατε στο ηφαίστειο και είπατε ότι το γεγονός αυτό πραγματικά ε, ήταν κάτι πολύ σημαντικό για το εξάμεινο αυτό. Κοιτάξτε, ναι, όντως, ε, δεν σας αποδίδω ευθύνε φυσικά για το ηφαίστειο, το αντίθετο μάλιστα, αλλά η κρίση του ηφαιστείου ήταν κάτι δυστυχές. Και ε, πραγματικά εδώ μας έδειξε ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός. Μας έδειξε την ανικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Και ε, κοιτάξτε, χωρίς να κατηγορώ κανένα, πρέπει να το διαπιστώνουμε αυτό, ότι υπήρξε ανικανότητα η Κομισιόν αντέδρασε κατόπιν όλης αυτής της κατάστασης και τελικά εντάξει νομίζω ότι είναι θετικά τα αποτελέσματα που προέκυψαν όμως παρέλυσε όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρέλυσαν τα κράτη, συγκλήθηκαν τα συμβούλια, ταχαίως θα έλεγα, πήραν τις κατάλληλες αποφάσεις όμως η αίσθηση αυτής της αδυναμίας ανάληψης δράσης ήταν τρομερή για όλους. Και έτσι λοιπόν ε, όλοι εξάγουμε το συμπέρασμα εδώ ότι πρέπει να παράξουμε περισσότερη Ευρώπη. Δεν μπορούν τα κράτη-μέλη να λαμβάνουν τις αποφάσεις μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά είδαμε ότι και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αναλάβει δράση, δεν έχει αυτή την ικανότητα. Έτσι λοιπόν, εντάξει, ας αφήσουμε το ηφαίστειο ως ένα γεγονός για να πούμε ότι ήταν ένα σοβαρό συμβάν το οποίο οδήγησε στο να λάβουμε κάποιες σημαντικές και σχετικές αποφάσεις. Τώρα, για τις μεταφορές, ε, ξέρετε, υπήρξε μια συμφωνία ε, για τις ενέργειες μεταφορές, πολύ σημαντική συμφωνία από πολιτική σκοπιά, η συμφωνία με τις Ηνωμένες σε σχέση με το δεύτερο στάδιο του ανοιχτού ουρανού μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΠΑ. Αυτή η συμφωνία αυτή είναι ε, μια συμφωνία που αφορά τις πτήσεις. Ε, είχαμε ε, τον κύριο Καγιέχα, όλοι θα τον γνωρίζετε, ο οποίος ε, πραγματικά εργάστηκε για την επίτευξη αυτής της συμφωνίας. Θέλω να το ποτίσω φόρο τιμής. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να αναγνωριστεί και στην Ισπανία, γιατί ίσως ε, στην Ισπανία δεν το γνωρίζουν. Τώρα, για το δίκτυο μεταφορών. Είχαμε τη συνεδρίαση στη Σαραγώσα, πολύ καλέ ήταν συζητήσεις και εγώ παρευρέθησα και ήταν ε, μια ευκαιρία να προβληματιστούμε για τις ικανότητές μας, για τι ανεπαρκίε μας, δεν μπορούσαν να ληφθούν εκεί οι αποφάσεις. Ε, εσείς ε, αρχικά όταν ήρθατε πρώτη φορά εδώ είπατε ότι δεν υπήρχε χρόνος ε, για να λάβετε αποφάσεις μέσα στο εξάμεινο, αλλά θα μπορούσαν να υιοθετηθούν κριτήρια. Ναι, υπάρχουν κριτήρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για τη λήψη αποφάσεων. Εδώ γνωρίζετε ότι έχουμε πάρα πολλές δυσκολίες, δεν μπορεί να συνεισφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση παραπάνω στο θέμα αυτό και ξέρετε ότι είναι και πάρα πολύ πολύ περιορισμένα τα κονδύλια των κρατών μελών. Όμως ε, όλα τα κράτη-μέλη θα κάνουν αυτές τις περικοπές. Έτσι λοιπόν έχουμε το πρόβλημα το ότι τα δίκτυα είναι ανεπαρκή. Αλλά κοιτάξτε, έχουμε συνεχεία περικοπές. Δηλαδή λέγαμε 20 δις στην αρχή, μετά 8 και τώρα τι συμβαίνει. Πρέπει να δούμε τι συμβαίνει. Δεν είχαμε χρόνο στη Σαραγώσα, αλλά ίσω κάποια στιγμή στην Επιτροπή αυτή θα έπρεπε να το συζητήσουμε αυτό το θέμα και με τα κρατη για να δούμε ποιο ε, διατίθεται να συνεισφέρει και να δούμε και ποια είναι και η πολιτική βούληση στα κράτη-μέλη για να συνεισφέρουν ε, το τμήμα των κονδυλίων που του αντιστοιχεί. Πρέπει να δούμε ποιο ε, είναι διατεθειμένο να συνεισφέρει και ποιο όχι και να δούμε ε, Ποιο μπορεί να υλοποιήσει αυτά τα νέα project όπως έχουμε το διάδρομο για τη Μεσόγειο να δούμε ποιος μπορεί να συνεισφέρει με πόρους και να δούμε αν μπορούμε να έχουμε ένα νέο ταμείο για τους πόρους αυτούς. Τώρα, θαλάσσιες μεταφορές. Συγγνώμη, πρέπει να τα πω γρήγορα γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, ούτε κι εσείς. Πάντω και σπανίς συνάδελφοι του κόμματό σας ε, σίγουρα ε, θα σας πούνε εδώ και θετικές κριτικέ, θα σας πούν θετικά πράγματα. Δεν χρειάζεται να τα πω εγώ. Λοιπόν, η ε, συμφωνία που υπεγράφει στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών ήταν πάρα πολύ χρήσιμη. Φαίνεται να είναι τεχνική, αλλά δεν είναι και τόσο τεχνική. Έχει μια μεγάλη πολιτική ε, σκοπιά και πραγματικά θα μας διευκολύνει στο να μειώσουμε τη γραφειοκρατία. Ουσιαστικά θα μπορέσουμε να επιλύσουμε κάποιες δυσκολίες ε, που έχουμε και ας μπούμε τώρα και στις συνδρομικές μεταφορές. Προσοχή εδώ όλοι επιδεικνύουν βούληση και θελοντισμό. Όμω η αλήθεια είναι ότι στι 24 Ιουνίου η Κομισιόν αποφάσισε να οδηγήσει, να προσφύγει στο δικαστήριο κατά 13 χαρών γιατί δεν είχαμε μεταφέρει σωστά την νομοθεσία του πρώτου πακέτου για τις συνδρομικές μεταφορές. Έτσι λοιπόν προσοχή εδώ γιατί πάρα πολλοί γνωρίζουν ότι πρέπει πέρα από τη βούληση να θέσουμε και πόρους, να χορηγήσουμε και πόρους. Και να τελειώσω. Δεν μπορούν ε, όλες οι προεδρίες ε, να υλοποιήσουν όλη τη δουλειά που είχαν θέσει ως στόχο από την αρχή. Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν έκλεισαν επαρκώς ε, και έχουμε και την έκθεση που θα πρέπει να κλείσει η Βελγική Προεδρία. Ε, εργαστήκατε εσείς σε κάποια θέματα, δεν μπόρεσατε να καταλήξετε σε συνένεση. Εγώ άσκησα κριτική για τα πολιτικά θέματα και το ξέρετε αυτό. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι όμως το τομέα αυτό έχετε εργαστεί επαρκώς, έτσι λοιπόν θα πω εντάξει δεν καλύψαμε όλους τους στόχους γιατί δεν είναι δυνατόν όμως ε, πραγματικά το αποτύπωμα που αφήσαμε είναι ενδιαφέρον. Και να σας πω ότι δεν μπορώ παρά να αναφέρω και τον κύριο Ορτής για τις θαλάσσιες μεταφορές, γιατί πραγματικά ε, εργάστηκε πάρα πολύ για το να κλείσει η έκθεση ΣΕΡ και υπήρχαν πάρα πολλές τεχνικές δυσκολίες, αλλά εγώ μπορώ να πω ότι τελικά καλά τα καταφέραμε. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ και συνεχίσουμε την ίδια οδό που ακολουθήσαμε και με το Μουντιάλ. Αν μας αφήσουν και οι υπόλοιποι βέβαια. Ευχαριστούμε, Πασκάλ. Ο Κύριος Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ θερμά για όλα όσα μα είπατε και κάνατε στην Προεδρία σα και για την άριστη συνεργασία που είχαμε από την αρχή μέχρι το τέλο της προεδρία. Όλοι είμαστε ικανοποιημένοι γι' αυτό. Αναφερθήκατε στο ειδικό πλαίσιο με στο οποίο χρειάστηκε να λειτουργήσει η οικονομική κρίση και όλα τα συναφή προβλήματα των μεταφορών και μετά η έκρηξη του ηφαιστείου που έδειξε ότι απαιτείται ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών. Θα πρέπει λοιπόν να ένσωμα, να ομαδοποιούμε τη δράση μας όσο πιο πολύ γίνεται και να συνεργαζόμαστε όσο περισσότερο. Αποκάλυψε πολλά αυτή η έκρηξη και θα χρειαστεί πολλή δουλειά τους επόμενους μήνες και χρόνια. Διότι αναφερθήκατε στο ενιαίο εναέριο χώρο, τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό που μιλάμε χρόνια και χρόνια και κατά κάποιο τρόπο επιταχύνθηκε η ολοκλήρωση του λόγου της κρίσης, ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να δούμε τι προθεσμίες πρέπει να τηρηθούν προκειμένου να πετύχουμε αυτόν τον ενιαίο ουρανό. Επίσης αναφερθήκατε στα δικαιώματα των επιβατών, πολύ σημαντικό για μας, γιατί υπάρχει χάσμα ανάμεσα στην νομοθεσία της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών στις αερομεταφορές και της πράξης. Υπάρχουν κενά και η Κομισιόν βέβαια θα κάνει προτάσεις να καλυφθούν αυτά τα κενά. Περνάω στους σιδηροδρόμους. Ακόμα σήμερα τα δίκτυα αυτά δεν είναι εναλλακτική λύση. Δέστε τι έγινε ας πούμε με την περίπτωση της έκρηξης του ηφαιστείου. Τι θέλω να πω στα, για τα τρένα πολλά μπορούν να γίνουν ακόμα για την σύνδεση των δικτύων, τις επενδύσεις κλπ. Συνολικά, αν ρίξουμε μια ματιά στον κατάλογο αυτόν που αναφέρεται, πολλά πράγματα έγιναν υπό την Προεδρία σας και δεν θα μπω στις λεπτομέρειες. Θα ήθελα μόνο να αναφέρω μερικά ενδεικτικά αναφερθήκατε στην τεχνολογία TS Intelligent Transport Systems οριστικοποιήθηκαν τα μέτρα αυτά κάτι λεπτομέρισμένο αυτές οι νέες τεχνολογίες γρήγορα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ένα πιο καθολικό τρόπο Είναι σημαντικό αυτό και για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, τις επιχειρήσεις σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Σε θέματα ασφάλειας υπάρχει ο κανονισμός για τα ατυχήματα και δυστυχήματα στις αερομεταφορές. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το μέτρο αυτό αν θέλουμε να αντιδρούμε γρήγορα και με άριστο τρόπο σε περίπτωση ενός δυστυχήματος. Μετά έχουμε την αποτελεσματική αποδοτική λειτουργία της ιστορικής αγοράς. Έχουμε την έκθεση STERX για το τι, ε, πώς πρέπει να διευκολύνονται διάφορες τυπικές διατυπώσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά τους εφοπλιστές. Άλλο σημαντικός κανονισμός για τις σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων. Με την εισαγωγή του One Stop Shop, ένα ενιαίο σημείο διαχείρισης που θα μας επιτρέπει με πιο αποτελεσματικό τρόπο να λειτουργούμε αν θέλουμε τα τρένα να είναι ανταγωνιστικά σε σχέση με τα άλλα μέσα μεταφοράς. Για τα δικαιώματα των ε, επιβατών αναφέρθηκα ήδη σε αερομεταφορές αλλά επειδή αναφερθήκατε και εσείς σε δύο άλλα μεγάλα θέματα μία έκθεση με την οποία ασχολήθηκε η συνάδελφος δίπλα μου για τα δικαιώματα των επιβατών στις ε, θαλάσσιες και πλωτές μεταφορές. Εδώ διαπιστώνουμε ευτυχώς ότι βρήκατε λύση. Αντίθετα δεν συμβαίνει το ίδιο και δεν προχωρήσετε πολύ για ένα άλλο μεγάλο θέμα που είναι τα δικαιώματα των επιβατών των λεωφορείων. Λεωφορεία Πούλμαν. Κάτι έχει ξεκινήσει, αλλά χρειάζεται δουλειά για τους επόμενους μήνες, προκειμένου να καταλήξουμε σε μια λύση με το Συμβούλιο. Τέλος, ένα άλλο σημαντικό σημείο, τα διευρωπαϊκά δίκτυα και οι σχετικές επενδύσεις. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο συνάδελφος Πασκουάλ για τη Σαραγώσα άριστα οργανωμένη συνάντηση αυτή και όλοι οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις θέσεις τους. Το Συμβούλιο, οι Κομισιόν, οι φορείς του κλάδου, μεγάλη ανταλλαγή απόψεων έγινε εκεί. Το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν έχουν ακριβώς τις ίδιες φιλοδοξίες νομίζω ως προς το πώς μπορούν να υλοποιηθούν αυτά τα διευρωπαϊκά δίκτυα όσο πιο γρήγορα και όσο πιο καλά γίνεται. Θα πρέπει να περιμένουμε τα πορίσματα προς το τέλος του χρόνου. Ένα όμως είναι σίγουρο. Όλοι συμφωνούμε ότι χρειάζεται δημιουργικό πνεύμα για να βρεθούν τα κονδύλια για να υλοποιηθούν όλα αυτά τα προγράμματα. Ο είναι αυτός που είναι, περιορισμένος. Πρέπει να δούμε τι άλλος τρόπος υπάρχει να βρεθούν χρήματα για να γίνουν αυτές οι αναγκαίες επενδύσεις για το ένα πραγματικά ενοποιημένο ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών. Και τώρα το πραγματικά τελευταίο θέμα, γιατί ήμουν εισηγητή στην πρώτη φάση. Βέβαια το Κοινοβούλιο ακόμα δεν έχει πάρει θέση για την συμφωνία αυτή με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Δεν έχει οριστικοποιηθεί η συμφωνία αυτή. Παραμένουν ακόμα ανισομέρειες στο μέτωπο αυτό. μα χάρη, οι Αμερικανικέ αεροπορικέ εταιρείε δεν τι μπορούν να κάνουν στην Ευρώπη σε σχέση με τι μπορούμε να κάνουμε εμεί στην Αμερική. Υπάρχει ανισομέρεια και πρέπει να λυθεί το πρόβλημα αυτό. Ωστόσο, κάποια προσέγγιση μεταξύ μα σημειώθηκε. Υπήρξε μια ε, ε οργάνων και από τις δύο πλευρές που συζητάει τα θέματα αυτά, όχι μόνο την πρόσβαση στην αγορά, την ασφάλεια, τη βιώσιμη μορφή μεταφορών, τα κοινωνικά, προκειμένου να υπάρξει μια προσέγγιση των δύο πλευρών για μια πιο ενοποιημένη υπερατλαντική αγορά. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ και πάλι θερμότητα για την άριστο πνεύμα συνεργασίας που επιδείξατε. Επαναλαμβάνω, πάρα πολλά κάνατε στην Προεδρία σας, πολλά επιτυχή. Δεν λύθηκαν όλα τα προβλήματα φυσικά. Πολλή δουλειά παραμένει ακόμα για τους διαδόχους σας, αλλά είναι φυσιολογικό. Μέσα σε λίγους μήνες δεν μπορεί κανείς να λύσει τέλεια τα πάντα. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπιλμπάου. Muchas gracias, presidente. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Υπουργό για το έργο του, το εξάμεινο αυτό. Και εμείς ε, θεωρήσαμε ότι κάνατε ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο γιατί έπρεπε να συμμετάσχουμε σε πολλούς φακέλους και να επιλύσουμε διάφορα προβλήματα. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα ήταν καλό παρόλα αυτά. Είναι αλήθεια ότι ήταν πολύπλοκη η Προεδρία και όχι μόνο έπρεπε να εργαστείτε στα πλαίσια μιας οικονομικής κρίσης ε, και στα πλαίσια της εικόνας που έδινε η Ισπανία προς τα έξω, αλλά αναφέρθηκε και το θέμα του ηφαιστείου. Εγώ συμφωνώ ότι ναι, οι κρίσεις πρέπει να μετατρέπονται σε ευκαιρίες για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον. Και θεωρώ ότι είναι ορθά τα συμπεράσματα τα οποία εξακάγατε. Όμως, προς την κατεύθυνση αυτή θα ήθελα να σας ρωτήσω. Πέρα από τις ε, συμφωνίες για τον Ευρωπαϊκό Ινέο Ουρανού, εδώ είδαμε ότι κάποια άτομα εθίγησαν ιδιαίτερα από την κρίση αυτή. Και θα ήθελα να σας πω ότι παρόλο που συμφωνώ με τις γενικές αρχές που αναφέρατε εσείς, να ρωτήσω αν γνωρίζουμε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα Δηλαδή, τι έγινε με τους χιλιάδες επιβάτες ε, που ζημιώθηκαν από την κρίση. Ανακοινώθηκαν κάποιες ε, κρατικές ενισχύσεις για τις εταιρείες και θα ήθελα να σας ρωτήσω μήπως μπορείτε να μας δώσετε κάποιες σχετικές πληροφορίες. Δηλαδή, τι έγινε με αυτές τις ενισχύσεις, ποια ήταν η διαχείριση, εγκρίθηκαν αυτές οι ενισχύσεις ή εγκρίθηκαν οι αποζημιώσεις για τους επιβάτες. Ο Επίτροπος ανακοίνωσε το ότι υπάρχουν τέτοιες κρατικές ενισχύσεις για τις εταιρείες. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να μας πείτε αν τελικά εγκρίθηκαν ή όχι, αν χορηγήθηκαν. Ποια, ποια ήταν η διαχείριση των αποζημιώσεων προς τους επιβάτες. Πώς τις διαχειρίστηκαν οι ευρωπαϊκές εταιρείες. Επίσης, σε ό,τι αφορά την προώθηση των σειρομικών διαδρόμων στη Σαραγώσα, θεώρησα ήταν σωστή η όθηση αυτή, τουλάχιστον από τα έγγραφα που μπόρεσα να διαβάσω, γιατί εγώ δεν μπορούσα να παρευρεθώ, αλλά βλέπω ότι προωθήθηκαν ε, τα έργα αυτά και η εκτέλεσή τους. Αλλά θα ήθελα να αναφερθώ το υπαριθμόν ε, τρία project. Σε μία από τις συμφωνίες λέγεται ότι θα γίνουν περαιτέρω προσπάθειες για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τα τμήματα που λείπουν εμπρόθεσμα για αυτό το project. Έτσι λοιπόν ρωτήσω αυτή η συμφωνία της Αραγώσα και οι προθεσμίες που έχουν προβλεφθεί θα γίνουν σεβαστές. Γιατί τουλάχιστον από όσα γνωρίζω εγώ ανακοινώθηκε ότι θα υπάρχει πιθανή μείωση του προϋπολογισμού και επομένως θα υπάρχει καθυστέρηση στην υλοποίηση αυτού του έργου, το οποίο αποτελεί προτεραιότητα. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να μου πείτε αν η δήλωση της Αραγώσα και άλλες ανακοινώσεις που έγιναν, αν συμπίπτουν ή αν αποκλίνουν. Επίσης να σας πω, πιστεύω ότι κάνατε πολύ μεγάλα προσπάθεια στην ακτή σε ό,τι αφορά του υδροδρομικούς διαδρόμους. Αλλά βάσει των συζητήσεων που είχαμε, σε ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, θεωρώ, δεν έχουμε ακόμη καθορίσει το ότι πρέπει και να έχουμε ξεκαθαρίσει ότι πρέπει να προωθούμε τα ευρωπαϊκά έργα. Από την προηγούμενη θητεία μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι δεν έχουν όλοι κατανοήσει με σαφήνεια ότι πρέπει να προσδιορίζουμε έργα που έχουν ευρωπαϊκή διάσταση. Πρέπει να καθορίζουμε τέτοια έργα και αναφέρομαι στην έκθεση Μαρινέσκος παράδειγμα. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή που είδαμε πραγματική κρίση στο φάκελο αυτό, έλαβε χώρα αυτή η κρίση γιατί δεν γνωρίζουν όλοι με σαφήνεια, ούτε στην Κομισιόν, ούτε στο Συμβούλιο, ούτε στο Κοινοβούλιο, ότι μια κρίση όπως αυτή του ηφαιστείου και όλος ο προβληματισμός σε σχέση με την αναγκαιότητα να προωθήσουμε αυτά τα ευρωπαϊκά project δεν είναι κάτι ξεκάθαρο. Και γενικά πρέπει να σας πω <laughs> ακόμη και αν προέρχεται από ε, το εθνικό ε, από το ΠΕΝΕΟΥΜΠΑ, από το Εθνικό Κόμμα των Βάσκων και είναι στην κυβέρνηση. Να σας πω ότι μία, ένα από τα πράγματα που έκανε η Ισπανική Προεδρία είναι που δεν, μάλλον που δεν έκανε είναι ότι θα έπρεπε να κάνουμε ένα προβληματισμό και να καταργήσουμε την εκπεριτροπή Προεδρία. Να έχουμε προεδρίες που πραγματικά να ηγούνται των ε, project και να προχωρούν με σαφήνεια σε όλα όσα έχουμε συμφωνήσει. Μπορεί να σας φαίνεται παράξενο αυτό, αλλά εγώ θα συνεχίσω να το λέω ότι δεν συμφωνώ με τις εκπεριτροπείς προεδρίες. Χρειαζόμαστε περισσότερη σταθερότητα. Χρειαζόμαστε καλύτερη ηγεσία. Χρειάζεται να καθορίσουμε μεγαλύτερη σαφήνεια τα ευρωπαϊκά project και να σας πω γενικά ότι Σωστά λέγονται τα πράγματα στις δηλώσεις, ασκείται κριτική στο ότι υπήρχε έλλειψη αντίδραση στην κρίση του ηφαιστείου. Γιατί εκείνη τη στιγμή, μέχρι που να περάσουν πέντε ημέρε, η Ευρώπη δεν ήξερε ποιοι είναι οι αρμόδιοι ευρωπαϊκοί θεσμοί για το θέμα αυτό και τι σκέφτονταν να κάνουν. Όμω, θεωρώ ότι τα συμπεράσματα που προέκυψαν στη συνέχεια είναι σωστά. Πρέπει να συνεχίσουμε να προχωρούμε προ την κατεύθυνση αυτή. Και επίση ε, υπήρξε και πρόοδο σε ό,τι αφορά γενικά τη βελτίωση των ε, δικαιωμάτων των επιβατών. Αν και έχουμε ένα κρεμμύ φάκελο για τους επιβάτες λεωφορείων. Και όπως σας είπα πρέπει να προωθήσουμε αυτά τα ευρωπαϊκά project. Και επίσης ε, άκουσα στην περίμεση σας αναφερθήκατε και σε αυτά τα σωματικά σκάνερ. Κοιτάξτε, για να μην θυμώσετε, να σας πω ότι εγώ είμαι υπέρ των σκάνερ γιατί πραγματικά έχω κουραστεί στα αεροδρόμια να με αγγίζουν παντού. Πραγματικά βαρέθηκα. Υπάρχουν και όρια. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να σε ψάχνει και να μην ξέρεις τι είναι θεμητό. Έτσι λοιπόν, με αυτά τα σκάνερ Σκέφτεστε να δώσετε μια προώθηση συνεργασία με την επόμενη Προεδρία. Έτσι λοιπόν να σας πω ότι σας ευχαριστώ για το έργο σας και θα ήθελα μεγαλύτερη ανάληψη δράσης στις στοιχές που αναφέρθηκα. Νομίζω δεν αναφερθήκατε στα θέματα αυτά στην παρέμβασή σας. Έτσι λοιπόν, αυτά στις στοιχές που ενδιαφέρουν τα μέλη της Επιτροπής να τις προωθήσουμε. Ευχαριστώ την κυρία Μπίλμπαου, ο κύριος Κράμερ. Σας παρακαλώ να με μακρηγορήσετε γιατί μάλλον θα χάσει και το μέσο μεταφοράς του υπουργό. Έχουμε ακόμη και έξι Έτσι λοιπόν θα ήθελα να σας παρακαλέσω να είστε σύντομοι. Ε, εντάξει, αλλά να έχουμε όλοι τα ίδια δικαιώματα. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιοι να μακρηγορούν και μετά εμείς να πρέπει να συντομεύουμε. Ε, σας ευχαριστούμε για αυτήν την ε, παρουσίαση και σας ευχαριστούμε για αυτή τη συνεργασία κύριε Υπουργέ. Έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν επανειλημμένα. Θα προσπαθήσω λοιπόν να εστιάσω σε κάποια ε, ζητήματα εδώ και θα περιοριστώ στις παρεμβασμού για άλλα. Σε ό,τι αφορά το ηφαίστειο θεωρώ πως ήταν πολύ σωστή απόφαση που ελήφθη δηλαδή να έχει απόλυτη προτεραιότητα η ασφάλεια των επιβατών. Για φανταστείτε εδώ ε, να, υπήρξε, να υπήρχε ένα αεροπλάνο το οποίο θα έπεφτε λόγω της ευαισθητικής λάβας τότε θα ε, συζητούσαμε πολύ διαφορετικά πράγματα τότε θα συζητούσαμε μόνο τα θύματα και ούτε οικονομικά ζητήματα ούτε οικονομίες ούτε τίποτα άλλο άρα λοιπόν ήταν πολύ σωστή η απόφαση που λήφθηκε τώρα σε ό,τι αφορά τους επιβάτες ε, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα τις ναυτιλιακές μεταφορές, δηλαδή τα καράβια, υπήρξαν εδώ συγκεκριμένες υποδομέ σε ό,τι αφορά τα άτομα με ειδικέ Αυτό δεν ισχύει για λεωφορεία, πράγμα που είναι πάρα πολύ λαθασμένο. Για παράδειγμα, ε, ε, μετά το Βιετνάμ ε, στι ΗΠΑ προβλέφθηκε ότι για όλα τα μέσα τη μεταφορά, δηλαδή και για τα λεωφορεία, να έχουν αυτέ τι υποδομέ για άτομα με αναπηρικό Ε, Θα πρέπει λοιπόν και εμεί να το επιβάλλουμε. Και εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με, τα μικρά λεωφορεία. Εδώ μιλάμε για τι μεγάλε επιχειρήσει λεωφορείων, οι οποίε μα είπαν ότι δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε κάτι τέτοιο. Είναι πολύ ε, ακριβό κάτι τέτοιο μιλάμε για το 30% των ανθρώπων οι οποίοι έχουν προβλήματα κινητικότητας. Ε, δηλαδή δεν μιλάμε μόνο για άτομα με αναπηρία, μιλάμε για ηλικιωμένου, μιλάμε για άτομα με ε, παιδικό καροτσάκι και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν αυτά τα άτομα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ε, αξιοποιήσουν τα μέσα μαζική μεταφορά. Ε, σε ό,τι αφορά την δήλωση τη Μαδρίτη και τον ε, κοινωνικό εναέριο χώρο, μα είπατε πω υπάρχουν κάποια πλεονεκτήματα. Ναι, το υποστηρίζω, αλλά μα είπατε ότι 5 ε, δισεκατομμύρια ευρώ εξοικονομούνται μέσω του ενιαίου εναέριου χώρου. Εάν το σκεφτόμαστε αυτό, τότε α σκεφτούμε πόσα μπορούμε να μειώσουμε κάποια ειδικότερα πλεονεκτήματα που προσφέρουμε. μόνο και μόνο λόγω της απαλλαγής από το ΦΠΑ και από τους ειδικούς φόρους για τα καύσιμα ε, λαμβάνει ουσιαστικά με, τη, με αυτή τη μορφή δηλαδή 30 δισεκατομμύρια ευρώ από τον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Λοιπόν, θα πρέπει να σταματήσουν αυτά τα προνόμια, αυτά τα πλεονεκτήματα. Μιλάμε για, μια, για ένα κλάδο ο οποίος πραγματικά είναι ε, ιδιαίτερα καταστροφικός για το περιβάλλον. Δεν μπορούμε λοιπόν να έχουμε ένα τέτοιο ε, δώρο, αν θέλετε, προς, την, ε, προς τις αεροπορικές εταιρείες, δηλαδή 30 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη Σαραγώσα και τους κοινού στόχους, είχαμε πει ναι, να εστιάσουμε στα bottlenecks, δηλαδή στα σημεία συμφόρησης και να υπάρχει και διευρωπαϊκή εμποδομένη, ναι, σε αυτό συμφωνήσαμε, αλλά ποιες είναι επιπτώσεις τελικά έχουμε 30 ε, ε, προτεραιότητες εδώ 20 ε, δισεκατομμύρια ζήτησε η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, τελικά 8 δισεκατομμύρια μας έδωσε το Συμβούλιο, τελικά τίποτα δεν έγινε, σε, δηλαδή ως περικοπές, τελικά είχαμε έγκριση για 9 διαδρόμους εδώ, corridors παρότι είχαμε προβλέψει αρχικά μόνο έξι. Άρα λοιπόν τι γίνεται με όλα αυτά. Δείχνει αυτό ότι δεν έχουμε τα απαραίτητα κονδύλια για να τα εφαρμόσουμε όλα αυτά. Ε, και αυτό σημαίνει με τη σειρά του ότι θα πρέπει να έχουμε μια διαφορετική πολιτική. Διαφορετική πολιτική για την κινητικότητα και από εκεί και μετά να δούμε ποια είναι τα κονδύλια που χρειαζόμαστε. Στη Σαραγώσα, ε, λοιπόν, εσεί είπατε, ε, δεν ξέρω αν συμφωνούσε και το Συμβούλιο ή όχι, πω ε, Ε, το κόστο ε, των υποδομών δεν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σε ό,τι αφορά τον υπολογισμό του δημοσιονομικού ελλείμματος. Ε, μα αυτό είναι, είναι καταστροφικό. Δηλαδή τότε δεν υπάρχει κανένα νόημα να, να, να θέτουμε ένα τέτοιο δημοσιονομικό έλλειμμα. Δηλαδή θα μπορεί να κάνει μια τέτοια ταχυτελεκτικά κόλπα ο κάθε υπουργό και να λέει αυτά τα έξοδα εγώ τα θεωρώ σε κόστο υποδομών και δεν θα υπάρχει καμία πίεση σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά δίκτυα. Έχουμε, έχουμε το Λιόν το τούνελ στις Άλπεις, ε, την ε, Μεσίνα και συνολικά τέσσερα τέτοια έργα υποδομής. και το κατά πόσο αυτά θα συγχρηματοδοτηθούν κατά 20, 30, 40% είναι ε, άσχετο. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να τα δούμε ολοκληρωμένα ε, όλα αυτά τα έργα, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια τη δική μα ζωή, αν και το εύχομαι. Αυτό λοιπόν που θα πρέπει να κάνουμε είναι να εστιάσουμε, να έχουμε συγκεκριμένε προτεραιότητε τι οποίε θα αρχίσουμε και αυτό θα πρέπει να επιτύχουμε και στο πνεύμα τη Αραγώσα. Ε, θα πρέπει λοιπόν να κατευθυνθούμε προς μια διαφορετική πολιτική. Μετά, κινητικότητα στις ε, πόλεις, αστική κινητικότητα. Και εδώ έχουμε να κάνουμε σημαντικό ζήτημα χρηματοδότησης. Το, στις από όλες το 70% όλων των ε, εκπομπών που είναι, βαρύνουν το περιβάλλον προέρχονται από την ε, κυκλοφορία των μέσων μεταφορών. Αλλά γνωρίζουμε ότι και στο 90% των ε, μετακινήσεων με αυτοκίνητο μέσα στις πόλεις είναι μικρότεροι από 6 χιλιόμετρα. Ναι, σωστά είπατε ότι θα πρέπει να εστιάσουμε στα μέσα μεταφορών. Αλλά εμείς ε, στην έκθεση Γκρόση μια πρόταση που είχαμε κάνει ότι να υπάρχει για παράδειγμα ένα σημαντικό ποσοστό 40% σε ό,τι αφορά ποδηλατόδρομους και ούτω καθεξής ε, και επένδυση μόνο κατά 20% στις, ε, στις, στους δρόμους απορρίφθηκε μια τέτοια προσέγγιση για παράδειγμα στη σημερινή κατάσταση όπως έχουμε το, το μεγαλύτερο ποσοστό κατευθύνεται προς την Στου ε, δρόμου, ε, του κανονικού και μόνο 0,9% κατευθύνεται για παράδειγμα προ την υποδομή για τους ποδηλατόδρομους. Άρα λοιπόν, ε, εδώ αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι διαφορετική αλλαγή σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότησή μα. Όμω μπλοκάρεται μια τέτοια αλλαγή τη πολιτική από το Συμβούλιο και γι' αυτό θα θέλαμε η Ισπανία να συμπαραταχθεί μαζί μα, δηλαδή να έχουμε πολύ μικρό ποσοστό σε ό,τι αφορά τι μεταφορέ στο, οχημάτων και να έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό χρηματοδότηση ε, για ε, του σιδηροδρόμου ε, και άλλα εναλλακτικά μέσα μεταφορά. Τώρα, εάν έχουμε, για παράδειγμα, ε, το πρώτο πακέτο για τους σιδηροδρόμους, ε, το οποίο τελικά ε, αντιμετωπίζει καθυστερήσεις και διαφοροποιήσεις μόνο και μόνο επειδή ο κύριος Μπαρόζο παρενέβη εκεί δεχόμενος πιέσεις από το Συμβούλιο, είναι κάτι που δεν μας βοηθάει. Είχαμε δηλαδή μια διαδικασία κατά παράβαση που είχε κινηθεί προηγούμενα και τώρα πάλι μια νέα καθυστέρηση. Εντάξει, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ε, το αν έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως τέτοια ε, νομική προσωπικότητα ή όχι, αλλά ε, σε κάθε περίπτωση δεν θα θέλουμε να υπάρχει η καταστατήγηση της κοινωτικής νομοθεσίας, γιατί αυτό που θέλουμε τελικά είναι καλύτερες μεταφορές στην Ευρώπη και καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Φώστερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να σας ε, συγχαρώ για τον ε, τελικό της ε, Κυριακής στην Ισπανία. Ο διαιτητής βέβαια δεν θα είναι πολύ ευπρόσδεκτος και σίγουρα δεν θα πάει για διακοπές στην Ολλανδία. Εν πάση περιπτώσει, συγχαρητήρια σε εσάς. Και τώρα, να σοβαρευτούμε να ευχαριστήσω τον Υπουργό. και όπως είπε ο συνάδελφός μας από το άλλο και είναι ευχάριστο ότι το βλέπουμε εδώ μαζί μας ενώπιον δηλαδή της Επιτροπής Μεταφόρους για τρίτη ή τέταρτη φορά κατά τη διάρκεια της Προεδρία του και ε, πραγματικά προσπάθησε η Ισπανική Προεδρία να προωθήσει ορισμένα ζητήματα τα οποία κρεμούν εδώ και αρκετά χρόνια. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ σε ορισμένα ζητήματα του, του κλάδου των αέριων μεταφορών. Καταρχήν σε ό,τι αφορά το ζήτημα της διερεύνησης ε, αντιχημάτων, θεωρώ πως ε, η Ισπανική Προεδρία και το Συμβούλιο έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο εδώ. Και όπως ξέρετε θα γίνει μια ακόμα συζήτηση το Σεπτέμβριο. Ε, σκοπεύουμε για πρώτη ανάγνωση εδώ. Πραγματικά θεωρούμε πως το Συμβούλιο έκανε μια πολύ καλή δουλειά προκειμένου να προσπαθήσει να βρει ένα συμβασμό στα ευαίσθητα ζητήματα και πραγματικά ε, ε, το προσωπικό από τι διάφορε επιδοτήσει για τη διαρρεύνηση αεροπορικών ατυχημάτων δείχνει να συμφωνεί με αυτή την προσέγγιση. Αναφερθήκατε επίση στο ζήτημα των ε, σαρωτών σώματο και πράγματι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήρθε εδώ και μα παρουσίασε ένα πολύ πλήρη φάκελο, τον οποίο καλωσορίζουμε. α, κάνω κι εγώ μια προσωπική παρατήρηση. Παρότι εγώ ανήκα προηγουμένως ε, στον κλάδο αυτό ε, δεν είμαι υπέρ ε, αυτής, αυτών των σαρωτών. Δηλαδή έχω ακόμα κάποιες ερωτήσεις εδώ. Θα ήθελα να, αξιοποιηθούν τεχνολογίες οι οποίες δεν χρησιμοποιούν ακτινοβολία και δεν χρησιμοποιούν την απεικόνιση του σώματος ενός προσώπου σε μια οθόνη. Δηλαδή κάτι τέτοιο ήδη έχει επιβληθεί ω υποχρεωτικό στο Ηνωμένο Βασίλειο, πράγμα που βέβαια μειώνει τι συζητήσει. Επίση θα πρέπει να υπάρχει μια πολύ καλύτερη ενημέρωση σε διασυνοριακό επίπεδο και ανταλλαγή των σχετικών ε, στοιχείων για έρευνε, ε, καλύτερη εξέταση των, ε, του, του προφίλ των επιβατών, ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πολύ σημαντικό πρόβλημα. Τώρα, ε, σε ό,τι αφορά την ε, συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών Open Skies ο Τσάντζο είναι πιο γνωστό στι ΗΠΑ από ότι ε, στην Ισπανία δεν ξέρω εγώ βέβαια είμαι από την Αγγλία αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που καταφέραμε πλέον με την σύναψη αυτής της συμφωνίας είναι ένα μεγάλο βήμα και εγώ θα ήθελα να επιστήσω ε, λίγο την προσοχή σε ό,τι αφορά ε, ε, την, τον έλεγχο των ξένων επενδύσεων, τον περιορισμό τους γιατί πραγματικά βλέπω εδώ να υποχωρούμε λίγο από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Quid pro είναι εδώ, έτσι, δηλαδή είναι μια ανταλλαγή, αν θέλετε. Και αυτό θα πρέπει να κάνουμε. Και ένα τελευταίο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω αφορά το Σέζαρ. είναι κρίμα που αξιοποιήσαμε την, ε, το ηφαίστειο και εκείνη την, ε, ε, εκείνο το ζήτημα και να προωθήσουμε το ΣΕΖΑΡ είναι πραγματικά πολύ σημαντικό και έχει διαρκέσει για πολλά χρόνια το ζήτημα αυτό. Είναι μεν περίπλοκο, αλλά πραγματικά θα πρέπει να το προωθήσουμε και μα άρεσε που είδαμε την Ισπανική Προεδρία να στείλει προ αυτή την κατεύθυνση. Γνωρίζουμε πω ο κλάδο έχει εργαστεί και έχει συνεργαστεί με το Κοινοβούλιο ε, για να το επιτύχει. Και ε, περνώ τώρα και στο Περσιακό έλεφο στη Στάχτη και το ζήτημα της, ε, των επιβατών. Κάποιοι πράγματι είχαν πολύ καλε μεταχείρισει και κάποιοι όχι. Αλλά κανένα δεν είχε φανταστεί ότι πραγματικά θα έκλεινε ο αέριο ε, ο χώρος για έξι μέρες ή περισσότερες αλλά, ε, μετά από την ε, τρομοκρατική επίθεση στις 10 Σεπτεμβρίου στην ε, Αμερική, όπου είχαμε πράγματι κλείσιμο του χώρου μεταξύ Ηνωμένου Βασιλού και Ηνωμένων Πολιτειών. Όμω τελικά το κόστο που προέκυψε από αυτό το κλείσιμο του ενέργου χώρου κόστησε 2 δισεκατομμύρια ευρώ για τα αεροδρόμια τη Ευρώπη. Και ε, υπήρξε μια πολύ καλή παρουσίαση, ε, ανακοίνωση από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το ζήτημα. Ε, και ε, είναι προφανέ ότι όλα τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα με του ε, προπολογισμού του και ειδικότερα η Ισπανική κυβέρνηση δεν έχει πολλά χρήματα εδώ να δαπανίσει. Οπότε υπάρχουν προβλήματα λοιπόν με τι αποζημιώσει, αλλά μιλάμε για πραγματικά αρκετέ μικρέ επιχειρήσει, όχι για τι μεγάλε αεροπορικέ εταιρείε που έχουν πληγεί από αυτό το κλεισμό. Ήταν πολύ καλή ομάδα της Ισπανικής Χωριδίας που εργάστηκε για αυτά τα ζητήματα. Ε, είμαστε όλοι ευχαριστημένοι με τις συζήτηση αυτές ε, που είχαμε και σας ευχόμαστε ό,τι ε, καλύτερο για το μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φώστερ. Μένουν τώρα πέντε ομιλητές, πέντε άτομα που έχουν ζητήσει το λόγο. Κύριος Υπουργός θα μπορέσει στη συνέχεια να σε απαντήσει και να γυρίσει σπίτι του. Λοιπόν, ε, νομίζω ότι όλες οι ομάδες έχουν τοποθετηθεί. Έτσι λοιπόν θα σας παρακαλούσα να είστε πιο σύντομοι. Ρος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εμεί ε, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε κύριε Υπουργέ για αυτή τη συνεργασία μα. Ε, είναι πολύ θετικό ο απολογισμός και για εμάς, για την Ευρώπη και για του πολίτες μας. Και θα ήθελα να συμφωνήσω με τα όσα είπε ο συνάδελφο από το ΕΛΚ, δηλαδή στον τομέα των ναυτιλιακών ε, μεταφορών αλλά και των αέριων ε, μεταφορών και το ζήτημα του ηφαιστείου. Πράγματι, ελήφθησαν σωστέ αποφάσει. Το ότι εντάξει δεν μπορούν να πετύχουν όλε τι προσπάθειε ε, που κάνουμε είναι γνωστό. Εντάξει, δεν το βιώσατε εσεί με τη δική σα ποδοσφαιρική ομάδα, το βιώσαμε εμεί, αλλά ποιο ξέρει στο, μέλλον μπορεί να στη δική μα ε, θέση. Από εκεί και μετά ε, θεωρώ πως σε κάποια ζητήματα υπάρχει υπερβολική αισιοδοξία και από την άλλη πλευρά ε, σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των επιβατών πραγματικά δεν υπάρχει πολύ θετική αντιμετώπιση από την πλευρά ορισμένων κρατών μελών. Μιλάω εδώ για τα λεωφορεία δηλαδή και στο γεγονό ότι οι επιβάτε πραγματικά θα ήθελαν να δουν περισσότερα από την πλευρά μα. Ε, και ειδικότερα σε σχέση και με τη συμφωνία με την Αμερική πω ε, και εκεί ε, δεν θα έπρεπε να είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι και σε σχέση με το SWIFT δηλαδή θα πρέπει να θυμίσουμε πω πρόκειται για διμερεί συμφωνίε, όχι μονομερείς ή μονόδρομες συμφωνίες. Δηλαδή έγιναν κάποιες δηλώσεις από την πλευρά τους αλλά καμία πρόθεση να, να λάβουν συγκεκριμένε αποφάσεις. Ε, σε ό,τι αφορά συντήματα χρηματοδότησης, ε, για παράδειγμα, να γίνουν κάποιες ε, επενδύσεις οι οποίες δεν σχετίζονται με σύμφωνο σταθερότητας και ούτω καθεξής, να πούμε ότι η δική σας αντιμετώπιση περιορίστηκε σε κάποιες δηλώσεις υποστηρικτικές, αλλά δεν είδαμε κάτι άλλο. Δηλαδή, είπαμε, είδαμε πολλά κράτη-μέλη τα οποία ε, ναι μεν δηλώνουν διατεθειμένα να προβούν σε περισσότερες δαπάνες αλλά τελικά δεν το πράττουν. Ε, και πραγματικά θα πρέπει να δημιουργηθεί μια γέφυρα μέτα ε, με τους διαρθρωτικούς ε, πόρους, ώστε να αξιοποιούνται ε, καλύτερα, όχι απλά να γίνονται περικοπές. Και καθώς η Ισπανία έχει να παίξει τη σημαντικό ρόλο, θα μπορούσε να βοηθήσει να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση μετά τη Σαραγώσα, ώστε να εφαρμοστεί στην πράξη. Κλείνοντας, σας εύχομαι μερικά ηφαίστεια ακόμα, ίσως και ένα ευρωπαϊκό ηφαίστειο. Ε, και ένα ηφαίστειο εσωτερικό αν θέλετε σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή βινιέτα και ένα ηφαίστειο και για τις χρηματοδοτήσεις γιατί υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη που βρίσκονται ακόμα μέσα σε μια τέτοια στάχτη. Γιατί πραγματικά μας έκανε τελικά καλό όλο αυτό το ζήτημα του ηφαίστειου. Ευχαριστώ. Έχουμε το Χαρούν Ταζιεύ της Κομισιόνα, ε. κυρία Αλβάρες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω για την αποτίμηση του έργου σας και για όλες τις δραστηριότητε που ανέλαβε το Υπουργείο. Κατά τη διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας, τόσο επί της ουσίας, όσο και σε ό,τι αφορά τους τύπους, νομίζω ότι κάνατε εδώ μια πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια να παρουσιαστείτε για να μας παρουσιάσετε τις εμπειρίες σας και να συζητήσουμε τα θέματα των μεταφορών. Πρόκειψε ένα θέμα που φαίνεται σημαντικό, το ανέφερε και ο κύριος Κράμερ και ο κύριος Γκρός, που είναι το θέμα της χρηματοδότησης. Και επίσης ε, ζητήθηκε να υπάρξει δημιουργικό πνεύμα για την ε, παροχή χρηματοδότησης. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να πω ότι ο κύριος Απατέρου μίλησε για δημιουργικό πνεύμα και ε, μάλιστα απάντησε σε μία αναφορά που έγινε στην Ισπανική ομάδα. Κάποιος ε, πρόβλεψε ότι πρόκειται να χάσουμε και ε, όμως η πραγματικότητα μας απέδειξε το αντίθετο. Και η κυρία Φοντένα μίλησε για διατησία. Ε, πάντοτε ο διαιτητή έχει ένα πολύ δύσκολο ρόλο, όμω εγώ δεν νομίζω ότι είμαστε και υπερβολικά ευχαριστημένοι, γιατί έτσι συμβαίνει στους διαφορούς αγώνες, όμως εγώ ήθελα να αναφερθώ στη χρηματοδότηση. Και στην περίπτωση αυτή στο ότι πρέπει να προσπαθούμε να άρουμε τα εμπόδια για να πετυχαίνουμε τους στόχους με διαφανή τρόπο. Έτσι εργάστηκε η Ισπανική Προεδρία, έτσι εργαστήκαμε και εμείς και έτσι ε, είδαμε και ότι και με το Μουντιάλ όταν θέτουμε κάποιους στόχους θέλουμε να κερδίζουμε. Έτσι λοιπόν πώς μπορούμε να το πράξουμε αυτό καταργώντας τα εμπόδια και ακολουθώντας την πορεία μας. Όμως εγώ νομίζω ότι ο Υπουργός έδωσε και ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα για το πώς πρέπει να διαχειριζόμαστε τις επενδύσεις στις ε, μεταφορές. Δεν πρέπει να έχουμε την ε, ίδια μεταχείριση της επενδύσεις αυτές ε, όπως σε άλλες περιπτώσεις. Και θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Γκρό ε, για την έκθεσή του, γιατί αναφέρθηκε στη χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση για μένα είναι κάτι ζωτική σημασία. Πρέπει να έχουμε δημιουργικό πνεύμα για να αναζητούμε μία λύσει, ε, λύσει όπω τέθηκε και από του υπόλοιπου συναδέλφου. Πρέπει να ακολουθήσουμε λοιπόν αυτή την οδό. Και αν μου επιτρέπετε, Προεδρία, καθώ έχω το λόγο, θα ήθελα να δράξω την ευκαιρία για να αποχαιρετήσω του συναδέλφου. Αυτή είναι η τελευταία μου παρέμβαση στο Κοινοβούλιο, γιατί την Παρασκευή θα αναλάβω καθηκόντα στο στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και θα ήθελα να σα ευχαριστήσω. Ε, με κάποιου συνεργάστηκα πιο στενά, με άλλου ε, είχα λιγότερη επαφή, αλλά όπω και να έχει θα ήθελα να σα ευχαριστήσω όλου. Ε, Κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και εγώ θα προσπαθήσω σύντομα να θίξω κάποια σημεία. Καταρχήν, να ξεκινήσω με τα δικαιώματα των επιβατών στα λεωφορεία. Ήμουνα εκεί ε, στον διάλογο μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων και πραγματικά ε, Λυπούμε που δεν φτάσαμε σε μια λύση. Δεν νομίζω πως είναι ευθύνη τη Ισπανία, νομίζω πως άλλοι ευθύνονται, αλλά είναι κρίμα πραγματικά γιατί είχαμε, ήμασταν πολύ κοντά σε μια λύση και ήθελα να είχαμε βρει μια λύση για του επιβάτε σε όλη την Ευρώπη. Τώρα βέβαια ε, θα πρέπει να πάμε στη διαδικασία ε, συνδιαλλαγή ε, που δεν είναι πάντα ό,τι καλύτερο. Εν πάση περιπτώσει θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ο κύριο Κρό είπε ότι θα ήθελα να είχαμε περισσότερα εφέστια. Νομίζω πω έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί το, αυτή, αυτό το, το γεγονό μα έδειξε πού ακριβώ υπάρχουν αδυναμίε στο δικό μα σύστημα. δηλαδή δεν ήμασταν προετοιμασμένοι και δεν μπορούσε να κάνει κάτι η Ισπανία και ε, πραγματικά δεν είμαστε προετοιμασμένοι όπω ε, άλλε περιοχέ ε, του πλανήτη, στι οποίε τα ηφαίστεια βρίσκονται στην μερίσια διάταξη. Και δεν ξέρω ε, ποιο ήταν από τα δύο πρώτο η εκείνη συνεδρία στην Ισπανία ή το ηφαίστειο, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, αυτή η περίπτωση του ηφαιστείου μας βοήθησε να προωθήσουμε ακόμα περισσότερο το νέο σύστημα κρατήσεων για του ε, σιδηροδρόμου ε, στην Ευρώπη. Ε, αυτό σχετίζεται και με τις προσπάθειες της Ισπανικής Προεδρίας και είναι πολύ θετικό. αγώσια αναφέρθηκα ήδη και ως εισηγήτρια σχετικής έκθεσης ε, σε ό,τι αφορά τα έργα, τα projects που προσπαθήσαμε να προωθήσουμε. Ε, έγιναν δυστυχώ κάποιε προτάσει ε, για το πώ θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε, αλλά δυστυχώ δεν είναι εύκολο να εφαρμοστούν τα πάντα. Προσπαθήσαμε να ιεραρχήσουμε κάποια project, να του δώσουμε προτεραιότητα, αλλά και αυτό ακόμα είναι δύσκολο. Από εκεί και μετά, ασφάλεια σε νέε μεταφορέ. Χαιρετίζω την, την πρώτη ανάγνωση που έγινε, γιατί πραγματικά είναι σημαντικό να γίνεται σωστά η διαρεύνηση των ατυχημάτων. Ε, τώρα σε ό,τι αφορά τους ε, σκάνες ε, προφανώς θα μας απασχολήσουν ακόμα περισσότερο. Μετά σε ό,τι αφορά τις, πώς τα καράβια πράγματι θα πρέπει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες και να αναφερθώ τέλος και σε κάτι στο οποίο δεν το οποίο δεν συζητήθηκε. Στην Κιχόν ε, έγινε η πρώτη, ε, υπήρξε η πρώτη μερίδα σε ό,τι αφορά τις ε, ευρωπαϊκές θάλασσες. Εγώ πραγματικά είδα πως είχατε μια πολύ καλά διοργανωμένη μερίδα εκεί. Δείχτηκαν πάρα πολλά ενδιαφέροντα ζητήματα. Σας ευχαριστώ λοιπόν και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για τις συμβαλλοντικές σας εργασίες. Η κυρία Λίχτεμπεργκ θέλει. Η κυρία Γιάλα Σέντερ τελευταία. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Υπουργό για τη διαθεσιμότητά του. Νομίζω ότι είστε ο Υπουργό που περισσότερε φορέ ήρθε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπω είχατε υποσχεθεί και από την αρχή. Και επίση, ε, ε, φυσικά να σα πω ότι όπω κερδίσαμε και το Μουντιάλ μέσω ομαδική δουλειά, ε, πιστεύω ότι και εδώ ε, και στη δική μας περίπτωση κάναμε πολύ καλή ομαδική δουλειά. Πραγματικά θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμής στην ομάδα σας και στη μόνιμη αντιπροσωπεία και νομίζω ότι και στο Υπουργείο είχατε πάρα πολύ καλή ομάδα και πραγματικά κατάλαβε ποιες είναι οι απαιτήσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μπορώ να σας πω ότι ε, και ο εκδημοκρατισμός των εργασιών μας ε, βοηθούν ε, σε αυτό. Επίσης, θα ήθελα να αναγνωρίσω την αδιάκοπη δουλειά του κυρίου Καγιέχα. Όμως, πολλά χρόνια είναι εδώ ο κύριος Καγιέχα και νομίζω όμως ότι του έλειπε να ασχοληθεί και με ένα διαφορετικό τομέα. Έτσι, λοιπόν, θα ήθελα να αφαιρθώ και στη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Πολιτείες ήμασταν ε, πάρα πολλά έτη τελματωμένοι σε κύκλους, σε γύρους συζητήσεων που ποτέ δεν έκλειναν. Ε, έτσι λοιπόν ε, αυτή τη φορά καταλήξαμε σε μια συμφωνία και αυτό χρησιμεύσε πάρα πολύ για στο να προωθηθούν σημαντικές πτυχές για την υλοποίηση του ανοικτού ουρανού αλλά φυσικά έδωσε και μία νέα δυναμική στον ενίο ευρωπαϊκό ουρανό. Επίσης θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συνεδρίαση της Αραγώσα. Καταλήξαμε σε μία συμφωνία με την Κομισιόν στη Σαραγώσα και αυτό μου επιτρέπει να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους γιατί υπήρξε μια πολύ μεγάλη αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκεί και έδειξε το πόσο ενδιαφέρεται αυτό το Κοινοβούλιο και πόσο δεσμεύεται για την υλοποίηση των δικτύων υποδομών και κυρίως ε, πρέπει να έχουμε μία εναλλακτική καθώς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα διέξοδο και το είδαμε αυτό και με την κρίση του εφεστίου. Πρέπει να έχουμε και ένα εναλλακτικό δίκτυο και ο σιδηρόδρομος πρέπει εκεί να διαδραματίζει τον κύριο ρόλο. Τώρα, για το θέμα του ενιαίου ουρανού, και ένα μνημόνιο στη Μαδρίτη από Πορτογαλία και Ισπανία και θα ήθελα να αναφερθώ εδώ σε αυτές τις δεσμεύσεις γιατί πολλές φορές εμείς ε, εδώ στο Κοινοβούλιο προχωρούμε αλλά δεν σημειώνουν πρόοδο τα κράτη-μέλη. Και στη Σέραγος υπεγράφησαν ορισμένα μνημόνια και ένα ε, πολύ σημαντικό το οποίο αναφέρεται στο Project 16 το κεντρικό άξονα και θα ήθελα να ζητήσω Ισπανία σε σχέση και με τις επόμενες δύο προεδρίες ε, να συμβάλλει έτσι ώστε να έχουμε τέτοια μνημόνια γιατί για αυτό το μνημόνιο μίλησαν και πάρα πολύ θετικά και αρμόδιοι υπουργοί από Πορτογαλία και Γαλλία. Έτσι λοιπόν είδαμε ότι δημιουργήθηκε μια δυναμική για τη δέσμευση των κρατών μελών. Όταν μιλάμε για δέσμευση, αλήθεια είναι, χρειαζόμαστε περισσότερους σπόρους, όμως ε, πρέπει να υπάρξει και δημιουργικό πνεύμα σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση από τα κράτη-μέλη. Αναφέρθηκε σε αυτό και η κυρία Άλβαρες πρέπει στο εσωτερικό των κρατών μελών να αναλυφθούν οι δεσμεύσεις και να υπάρχει δυναμική έτσι ώστε και η Ευρωπαϊκή Ένωση να κατορθώσει να συστήσει ένα φιλόδοξο ταμείο για τις υποδομές και για τη μεταφορά. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί στο τελευταίο Συμβούλιο μιλήσατε για το σημαντικό ρόλο που έχουν οι μεταφορές στρατηγική το 2020. Ο ε, κύριος Κάλλας ε, το ίσως για την τελευταία στιγμή, όμως το ότι η Ισπανική Προεδρία έβαλε αυτή τη συμπληρωματική πτυχή ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Και εγώ θα ήθελα να σας ζητήσω, εσείς ως αρμόδιο υπουργό να συνσφέρετε κάθε φορά έτσι ώστε να επισέρχεται αυτό το στοιχείο στη συζήτηση για τις δημοσιονομικές προοπτικές. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω την Προεδρία για όλο το έργο της, γιατί έκλεισε το φάκελο των δικαιωμάτων των επιβατών στι θαλάσσιε μεταφορέ. εξαιρετική δουλειά και επίσης ε, για τα δικαιώματα των ε, ατόμων με ειδικέ ανάγκες. Μας ευχαρίστησε ε, η οργάνωση των ατόμων αυτών. Τώρα βέβαια για το φάκελο των μεταφορών με λεωφορείο ελπίζω εσείς ως υπουργό να βοηθήσετε την επόμενη Προεδρία να καταλήξει σε συμβασμό για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Να δώσουμε τώρα τον λόγο στον κύριο Υπουργό. Και φυσικά να τον ευχαριστήσουμε και για την ε, παρουσία του σήμερα εδώ, αλλά και για την ε, μεγάλη διαθεσιμότητά του καθ' όλη την Προεδρία. Η κυρία Σάντερς ε, το είπε ότι ήταν ο υπουργό που ήρθε περισσότερες φορές εδώ στο Κοινοβούλιο επειδή ξέρετε ε, ότι και με την ε, κρίση, ε, με το ηφαίστειο που μακρινθήκαμε πολλές φορές από τα εθνικά προβλήματα και είδαμε ότι ήταν διεθνείς οι κρίσεις πολλές φορές. Πολλά έγιναν, το υπενθυμίσατε βέβαια, υπήρξαν και κάποιες δράσεις που δεν μπόρεσαν να ελοπιθούν, δεν υπήρξε ευκαιρία, δεν υπήρξε και χρόνος, δεν μας επέτρεψαν οι συνθήκες. Οι συνθήκες να υλοποιηθούν όλε οι δράσει, όμω ήταν πολύ καλή η Προεδρία. Σα σας ξαναδώσω το λόγο, κύριε Υπουργέ, για να απαντήσετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους κυρίους ε, βουλευτές για τα ευγενικά τους λόγια, καθώς αναγνώρισαν το έργο που υλοποιήθηκε κατά την Ισπανική Προεδρία στο θέμα των μεταφορών. Θέλω να ευχαριστήσω κυρίως ε, και όσα είπαν ε, κύριε Λεγκράντ και σας Μπιλμπάου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το ότι ε, δώσατε έμφαση επίσης σε όλα τα εκρεμή ζητήματα, δηλαδή για τους στόχους και τις προκλήσεις ε, που εξακολουθούν να παραμένουν εκρεμή και σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Το είπα και στην παρέμβασή μου και θέλω να το επαναλάβω. Εγώ πραγματικά αισθάνθηκα ότι ε, το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της παιδείας διαδραμάτισε ένα καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη πολλών συμφωνιών, κυρίως την επίτευξη της συμφωνίας με τη ΣΥΠΑ. πρόεδρος της Επιτροπής ε, Μεταφορών, αλλά ε, και η Κομισιόν ε, και η Κορεπέρ συμμετείχαν τα μάλλον, αναφέρθηκαν εδώ διάφοροι συνάδελφοι και κυρίως Καγιέχα. Όλοι είχαν την δυνατότητα να συνεισφέρουν προσωπικά και θα ήθελα να το τονίσω αυτό επίσης. Ήταν μια ομαδική δουλειά εμείς θέταμε κοινού στόχους για να πετύχουμε τις προκλήσεις που είχαμε θέσει. Τώρα, θα ήθελα να κάνω και μία συμπλήρωση στην αρχική μου παρέμβαση και θα ξεκινήσω με το ηφαίστειο. Σας ευχαριστώ τα όσα είπατε για τη διαχείριση της κρίσης ε, του ηφαιστείου, όμως είναι αλήθεια ότι πραγματικά παρουσιάστηκαν εμφανώς και οι λήψεις που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να απαντήσει σε προκλήσεις που εκδηλώθηκαν σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, το είχα πει αυτό και την πρώτη φορά ε, που παρευρέθηκα εδώ, ότι είχαμε ενίο νόμισμα, αλλά δεν έχουμε ενίο ουρανό. Και αυτό το είδαμε ξεκάθαρα με την κρίση του εφεστίου. Όμως είναι αλήθεια ότι από την πρώτη μέρα, όχι την πέμπτη μέρα, από την πρώτη μέρα ενεργοποίησαμε το Ευρωκοντρόλ, ενεργοποίησαμε τους συντονιστικούς μηχανισμούς με την Κομισιόν και επίσης διμερώς με τα κράτη-μέλη. Γιατί Ας μην ξεχνάμε ότι η ικανότητα λήψης αποφάσεων ε, ήταν των κρατών μελών. Την αρμοδιότητα την είχαν τα κράτη-μέλη πέρα από το ότι ε, υπήρξαν κοινά ζητήματα που εκδηλώθηκαν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως η διαχείριση αυτή μας ε, έδειξε το ότι πρέπει να ενισχυθούν ορισμένες ε, πτυχές ανάληψης πρωτοβουλειών έτσι ώστε στο μέλλον να μπορούμε να έχουμε μια πιο αποτελεσματική και ευέλικτη διαχείριση και ταυτόχρονα να μπορούμε να έχουμε μικρότερο στον εναέριο χώρο. Κάναμε, σημειώσαμε αρκετή πρόοδο, δεν θα ήθελα να τα ξαναπώ. Προωθήσαμε την εφαρμογή του ενεωρανού και επίσης όλα τα κρατημέλη συνειδητοποίησαν ότι έπρεπε να υιοθετηθούν ορισμένα μέτρα. Όμως πιστέψαμε ότι όταν εγώ κάλεσα το έκτακτο συμβούλιο των Υπουργών, μεταφορών, πραγματικά ε, εγώ αισθάνθηκα πολύ περίεργα ε, γιατί ε, ενώ ήταν εθνικές οι αρμοδιότητες έπρεπε να ληφθούν κάποιες αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο όμως οι αποφάσει αυτέ έπρεπε να ληφθούν έτσι ώστε να εγγυηθούμε σε κάθε περίπτωση την ασφάλεια. Γιατί δεν γνωρίζαμε σε πολλέ περιπτώσει πώ αυτά τα σηματίδια ε, ουσιαστικά τι επίπτωση είχαν στι μηχανέ των αεροσκαφών. Και έπρεπε τελικά να αποφύγουμε να λάβουμε κάποιες βιαστικές αποφάσεις. Ε, κάποιος είπε ότι δεν είχαμε λάβει βιαστική απόφαση και είχαμε οδυνηρές συνέπειες. Ε, σήμερα θα μιλούσαμε διαφορετικά για το θέμα. Όμως ε, η έκρηξη του ηφαιστείου ανέδειξε και άλλο ζήτημα την αδυναμία της επικοινωνίας στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να προωθήσουμε τα διευρωπαϊκά δίκτυα, κυρίως τα σιδηροδρομικά. Λοιπόν, έχουμε σιδηροδρομικά δίκτυα ως εναλλακτική για τις ενέργειες μεταφορές. Και σε σχέση με αυτό να πω ότι όταν ε, ε, κάποιοι ευρωβουλευτές αναφέρθηκαν στην ε, αναγκαιότητα οι επενδύσεις στα διευρωπαϊκά δίκτυα και δεν αναφέρομαι στο σύνολο των υποδομών, περιορίζομαι στα διευρωπαϊκά δίκτυα που είναι κάτι με το οποίο συμφωνούν όλα ε, τα κράτη-μέλη και χρησιμοποιούν όλα τα κράτη-μέλη, να σας πω ότι οι επενδύσεις των ίδιων των κρατών μελών ε, πρέπει να ε, δίνονται τη στιγμή που θέτουμε προτεραιότητα στο δίκτυο των μεταφορών. Όμως, εδώ θέλουμε ουσιαστικά να προωθήσουμε τις επενδύσεις και σε επίπεδο κρατομελών, γιατί Κοιτάξτε, πρόκειται για ευρωπαϊκά δίκτυα. Δεν εποφελούνται μόνο ορισμένα κράτη-μέλη από αυτό. Πρέπει να δημιουργήσουμε συμπληρωματικούς μηχανισμούς χρηματοδότησης πέρα από τους πόρους που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί. Και συζητήσαμε και το ρόλο που μπορεί να έχουν οι ΣΔΙΤ, κυρίως στην ανάπτυξη είδων υποδομών αλλά η ίδια η Κομισιόν, ο ίδιος ο Επίτροπος και τα κράτη-μέλη γνωρίζουν ότι αν δεν είμαστε ικανοί να δημιουργήσουμε μηχανισμούς χρηματοδότησης για τις υποδομές σιδηρομικών μεταφορών, δεν θα είμαστε σε θέση να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει. Ε, έγινε μια αναφορά από την κυρία Βιλμπάου στο στην Ισπανική δέσμευση για το διάδρομο 3 και για το διάδρομο 16 γιατί αυτή ήταν ε, ακριβώς ε, το αντικείμενο της υπογραφής ενός μνημονίου μεταξύ Ισπανίας, Γαλλίας και Πορτογαλίας για να συνεχίσουμε να δηλώνουμε το στρατηγικό χαρακτήρα αυτών των διαδρόμων. Μάλιστα αναφέρθηκε και στην εθνική πολιτική και θέλω να απαντήσω σε αυτό. Η προτεραιότητα του Υπουργείου ε, για τις δημόσιες ε, υποδομές είναι να συνεχίσει να προωθεί τις ιδρομικές μεταφορές και φυσικά θέλουμε να προωθήσουμε το δίκτυο για τα εμπορεύματα, το δίκτυο για τους επιβάτες, τις ε, τοπικές μεταφορές και την υψηλή ταχύτητα φυσικά στα δίκτυα προτεραιότητας εντάσσονται και οι στόχοι που έχουμε για τις αεροδρομικές μεταφορές. Έτσι λοιπόν, εδώ δεν ξαναθέτω προς αναθεώρηση κανένα χρονοδιάγραμμα για τις ημερομηνία της επίτευξης που έχουμε για τους άξιους προτεραιότητας. Φυσικά αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται τις δράσεις των υπολείπων κρατών ε, μελών. Έτσι λοιπόν ε, είχαμε και μια συνεδρίαση πολύ με τον κύριο Μπουσερό, τον συνάδελφο, τον Γάλλο συνάδελφο, για να προωθήσουμε το στόχο αυτό και κύριος θα γίνει στην διμερή διάσκεψη που θα λάβει χώρα το τελευταίο τρίμηνο του 2010. Έγινε και μία αναφορά στην ε, συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξέρετε ότι τη συμφωνία αυτή την διαπραγματευόμασταν το 2007. Είχαμε πάρα πολλές δυσκολίες και πραγματικά εκεί σημειώθηκε σημαντική πρόοδος. Μπορούμε να έχουμε περισσότερες ε, φιλοδοξίες. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε ξεκινήσει μία διαδικασία που θα επιτρέψει την απελευθέρωση θα επιτρέψει τις αμοιβέ επενδύσεις, να μειώσουμε τις αποστάσεις και φυσικά όλα αυτά θα έχουν πολύ σημαντικό αντίκτυπο και στις ε, εκπομπές των αερίων. Αλλά όπως σας είπα θα υπάρχουν και αμοιβέ επενδύσεις και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι λοιπόν μια συμφωνία που θα μπορούσε να πάει πιο πέρα, αλλά ήδη έχουν τεθεί οι βάσεις μιας ήδη προηγμένη διαδικασία. Και πρέπει να συνεχίσουμε φυσικά να εργαζόμαστε στον τομέα αυτό, γιατί πρέπει να εκπονήσουμε και νομοθεσία για να μπορέσουμε αμοιβαία να προβούμε στην απελευθέρωση του καθεστώτος επενδύσεων. Αναφέρθηκα στη συνάντηση της Αραγώσα. Ε, γενικά, να σας πω ότι εγώ θεωρώ πολύ θετικό τον όλο προβληματισμό που υλοποιήθηκε, όμως ε, φυσικά Καθώς είμαι υπουργό ενό κράτου μέλου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, αρμόδιο για τα θέματα αυτά, συμφωνώ ακόμη περισσότερο και πρέπει να αναζητήσουμε εναλλακτικού πόρου για να συνεχίσουμε να προφούμε τι επενδύσει στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών. Λοιπόν, ε, σε ό,τι αφορά τώρα τις ε, διατυπώσεις ενημέρωσης για τα σκάφη, αυτό αποτελεί πάρα πολύ σημαντικό βήμα για το να δημιουργήσουμε έναν Ευρωπαίο θαλάσσιο χώρο χωρίς σύνορα και αυτό φυσικά σημαίνει ότι θα μειωθεί το κόστος των προϊόντων που μεταφέρονται και θα μειωθεί ε, η χρήση των οδικών οδών προχωρήσαμε με τον ίδιο τρόπο. Νομίζω ότι αναφέρθηκαν σε αυτό... Ε, αναφέρθηκε σε αυτό ο κύριος Δεγκράντη για το σιδηροδρομικό πακέτο, όμω στο πλαίσιο του προγράμματος του Τρίου των Προεδριών θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τη Βελγική Προεδρία για να προωθήσουμε την αθεώρηση του πρώτου πακέτου για του σιδηροδρόμου με κύριο στοιχείο τη βελτίωση και διευκόλυνση των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα αναφερθώ τώρα στο, στο θέμα της, ε, ε, των ατυχημάτων στις ενέργειες μεταφορές. Θεωρώ ότι πετύχαμε κάποιο θετικό αποτέλεσμα και λυπάμαι που δεν μπορούσαμε να ελοπίσουμε μια συμφωνία για τα δικαιώματα των επιβατών για τα λεωφορεία που μετακινούνται με λεωφορεία. Είχαμε φτάσει ε, σε ένα σημείο κοντά στην επίτευξη. Ελπίζω να πετύχουμε τη συμφωνία αυτή υπό τη Βελική Προεδρία. Είναι προτεραιότητα και φυσικά θα συνεχίσω να ασκώ πίεση προς αυτήν την κατεύθυνση με Βέλγο συνάδελφο. Σαν να ήμουν εγώ πρόεδρος ε, του Συμβουλίου Μεταφορών θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να πετύχουμε τη συμφωνία αυτή. Αναφερθήκατε και στην αστική κινητικότητα. Εγώ νομίζω ότι τα συμπεράσματα της συνεδρίας της Ακορούνια υποστηρίζουν την λήψη συγκεκριμένων μέτρων για να υποστηρίξουμε την αηφόρο κινητικότητα, όπως ε, να προωθήσουμε τη λογική χρήση του γιοταχή και να προωθήσουμε τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς, να βελτιώσουμε την εφοδιαστική για τη μεταφορά των εμπερευμάτων, να προωθήσουμε νέες τεχνολογίες για οχήματα, για καύσιμα, να βελτιώσουμε την οδική ασφάλεια, να προωθήσουμε τη χρήση του ηλεκτρικού αυτοκινήτου στις πόλεις, στις αστικές περιοχές. Είναι σημαντικά αυτά τα συμπεράσματα και τώρα πρέπει να τα αναπτύξουμε, αλλά έχουμε ήδη ένα πλαίσιο προβληματισμού με το οποίο όλοι συμφωνούμε και το οποίο βρίσκει σύμφωνα όλα τα κράτη-μέλη και αυτό έγινε προφανές με την επικύρωση των συμπερασμάτων στο Συμβούλιο Μεταφορών σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό αυτοκόλλητο, το Ευρωβινιέτ, ευρωπαϊκό σήμα. Ε, μπορώ να σας πω ότι στις 27 Ιανουαρίου εγώ παρευρέθησα στην Αρμόδια εδώ και τον Ιούνιο είχαμε μια τεχνική συνεδρίαση για να συζητήσουμε την αντίκτυπο της εφαρμογής αυτής της οδηγίας που υλοποιεί κομπισιόν μέσω του Ινστιτούτου Τεχνολογικών Προοπτικών και ζητήσαμε από την Κομισιόν μία επικαιροποίηση για τα αποτελέσματα της εφαρμογής της σημερινής οδηγίας για αυτό το ευρωπαϊκό σήμα για να προσπαθήσουμε να δούμε ποιες είναι οι εμπειρίες των κρατών μελών για ε, την τιμολόγηση των βαρέων οχημάτων. Η οδηγία αυτή αναμφισβήτητα στο μέλλον ε, θα χρησιμοποιηθεί ε, με κατάλληλο τρόπο, όμως για να γίνει αυτό πρέπει να διασκεδάσουμε τις αμφιβολίες που υπάρχουν ήδη επί της οδηγίας αυτής. Και αυτό αποτελεί έναν από τους στόχους που έχουν τεθεί ήδη στη Βελγική Προεδρία και φυσικά η Ισπανία θα συμμετάσχει. Κυρίες και κύριοι, με αυτές τις σκέψεις γενικού χαρακτήρα θεωρώ ότι ολοκληρώνω εδώ την παρέμβασή μου σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας. Σας ευχαριστώ για τα όσα είπατε σήμερα, για το έργο που υλοποιήσαμε. Έχουμε πάρα πολλούς κοινού στόχους, πάρα πολλές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και είμαι σίγουρος ότι με κοινή δουλειά και με αφοσίωση και με αυτό το ομαδικό πνεύμα το οποίο διέπει τον τρόπο εργασίας αυτής της Επιτροπής, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και έτσι θα προωθήσουμε την επίτευξη των στόχων αυτών και να σας πω ότι πάντοτε θα έχετε τη δική μου συνεργασία. Σας ευχαριστώ πολύ.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 allons maintenant parler de l'accord entre la communauté européenne et le canada sur la sécurité de l'aviation civile. Η Πρώτη αεροπορική συμφωνία για την Λισαβόνα. Το στην Κομισιόν. και μετά θα ακολουθήσει η συζήτηση. Thank you very much, Mr. President. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να σας αναφέρω για τη συμφωνία αυτή με τον Καναδά. Δύο συμφωνίες είναι. Η η συνολική πλήρης συμφωνία για την αεροπορική ασφάλεια με υψηλή σύγκληση στα θέματα αυτά και απελευθέρωση επίσης και μια δεύτερη συμφωνία για την απελευθέρωση αεροπορικές υπηρεσίες στην υπερατλαντική αγορά με τη δεύτερη συμφωνία Ένωση ΗΠΑ. Αλλά όπως είπατε και εσείς έχουμε και τη συμφωνία για την ασφάλεια με σημαντικά ωφέλη με την αμοιβαία αναγνώριση από τον κλάδο και στην Ευρώπη και στον Καναδά. Γιατί οι συμπορικέ μα σχέσει αυτό είναι όλο και πιο σημαντικό σχέση με τον Καναδά και αυτή η συμφωνία θα δημιουργήσει και θέσει απασχόληση και θα μειώσει και τη γραφειοκρατία. Και θα μα ε, βοηθήσει στο να έχουμε μια ομαλή συνεργασία μεταξύ των εθνικών διοικήσεων. Η αγορά τη Ένωση και του Καναδά είναι πάνω από το 25% τη συνολική αγορά και οι οργανώσεις κατασκευή κινητήρων αεροπλάνων θα αφοληθούν πολύ από τη συμφωνία αυτή και πρόκειται για πρωταγωνιστές στον κόσμο. Οι συνδυασμένε εξαγωγές είναι πάνω από, γύρω πάνω από 50 δι και σε θέματα αεροδιαστημικής με κατασκευή ε, μιλάμε για 49 δις δισεκατομμύρια παραγωγή. Η ασφάλεια στον Βόρειο και Νότιο Ατλαντικό θα ωφεληθεί από τη συνεργασία αυτή μεταξύ Καναδά και ένωση. Όπως ξέρετε, παρόμοια συμφωνία ασφάλεια με τι ΗΠΑ υπάρχει ήδη, όπου να θα ολοκληρωθεί. Περιμένουμε την απάντηση του Κογκρέσου και αύριο στη διάσκεψη Ένωση Βραζιλία ο πρόεδρος Μπαρόσο θα υπογράψει τη συμφωνία με τη Βραζιλία. Πάντα για θέματα ασφάλειας στις αερομεταφορές. Μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ που θα εξοικονομούνται κάθε χρόνο χάρη σε πιο, στην έγκριση, πιο απλή έγκριση παραγωγής προϊόντων, αμοιβαία αναγνώριση. Οι αεροπορικέ εταιρείε θα ωφεληθούν επίσης γιατί υπάρχουν ειδικέ διατάξεις για την αμοιβαία χρήση εγκαταστάσεων για συντήρηση κλπ. Οι πολίτε θα ωφεληθούν από τα θέματα αυτά ασφάλεια. Το πιο σημαντικό, βέβαια, θα στηριχθούμε στην κοινωνία αυτή, στην συμφωνία αυτή, γιατί όπω ξέρετε, ο Ευρωπαϊκό Φορέα τη δόθηκε ε, ε, επιπλέον εντολή για τι άδειε των πιλότων κλπ. Και προετοιμάζεται το έδαφο για τη νέα αυτή δράση που θα στηριχτεί στη συμφωνία αυτή, προκειμένου να βρεθούν λύσεις και για τις αεροπορικές εταιρείες και για τα πληρώματα. Όντως είναι η πρώτη συμφωνία που θα καλυφθεί πλήρως από τη, συμφωνία, από τη συνθήκη της Λισαβόνας, ομόφωνη υποστήριξη όλων των υπουργών στο Συμβούλιο. Η καναδική πλευρά ήδη επικύρωσε τη συμφωνία και είπε κάτω κοινοποίηση αυτό στην Ένωση στις 30 Απριλίου. μεγάλες προσδοκίες να οριστικοποιηθούν και τυπικά να οριστικοποιηθεί μάλλον αυτή η συμφωνία και να αρχίσει η πρακτική της εφαρμογή. Όπως σας είπα αυτή η συμφωνία για την ασφάλεια συμπληρώνεται με την άλλη γενική συμφωνία με τον Καναδά που είναι πιο ευρία φυσικά γιατί καλύπτει ευρύς τομείς συνεργασίας και την πρώτη αυτή συμφωνία και εκεί θέλουμε την συνένεση του Ευρωκοινοβουλίου για να την προωθήσουμε. Και είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν η συγκεκριά μας η κυρία Τικάου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο, του εκπροσώπου μόνο της Κομισιόν γιατί πρόσφατα έγινε μια συνάντηση μεταξύ μας για να, να συζητήσουμε αυτές τις δύο συμφωνίες. Είναι δύο χωριστές συμφωνίες. Η Γενική Συμφωνία για τους κοινού... κοινούς κανόνες για θέματα ασφάλειας στην πολιτική αεροπορία. Σύντομα το Κοινοβούλιο θα πάρει ένα κείμενο από την Κομισιόν, το τελικό κείμενο εννοώ. Όλες οι κυβερνήσεις βέβαια θα πρέπει να επικυρώσουν τη συμφωνία. Αυτό χρειάζεται χρόνο. Τώρα, η συμφωνία μεταξύ της Ένωσης και του Καναδά πάλι για θέματα ασφάλειας με βάση μια απόφαση του ECJ για την άρση τεχνικών εμποδίων για το εμπόριο προϊόντων. Αυτό υπάγεται στην κοινή εμπορική πολιτική. Έχουμε λοιπόν αποκλειστική αρμοδιότητα για την Ένωση. Γι' αυτό για τη συμφωνία αυτή για την ασφάλεια στην πολιτική αεροπορία δεν χρειάζεται επικύρωση από όλα τα κράτη-μέλη. Απλώς χρειάζεται το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εγκρίνουν. Το Κοινοβούλιο θα γνωμοδοτήσει με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας μέχρι τώρα έξι χώρες μέλη έχουν κλείσει συμφωνίες με τον Καναδά διμερός. για την ασφάλεια στην πολιτική αεροπορία. Βέβαια όλες αυτές οι συμφωνίες ε, καταπίπτουν ε, καθίστανται περιττές από την επιθεσχή Νέα Συμφωνία Ένωσης Καναδά. Υπάρχει όμως μια σημαντική διαφορά μεταξύ των, διμερών, των έξι διμερών συμφωνιών και της νέας συμφωνίας. Στις ε, διαδικασίες εφαρμογής. Αυτές οι διαδικασίες εφαρμογής αυτή τη στιγμή είναι υποχρεωτικές, ενώ στη συμφωνία θα μπουν ως παραρτήματα. με νομική ισχύ. Αυτό είναι το νέο στοιχείο. Πιο πριν οι διατάξεις αυτές άρχισαν να ισχύουν μόνο αν υπήρχαν νέες διμερείς συμφωνίες μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών μεταξύ του Καναδά και της συγκεκριμένη χώρας μέλους. Τώρα, οι εφαρμοστικές αυτές διατάξεις θα έχουν νομική ισχύ είναι αναπόσπαστο κομμάτι της συμφωνίας και είναι και υποχρεωτικές. Με τον κανονισμό 1592 του 2002 για τη σύσταση της ESA που αργότερα αντικαταστάθηκε με τον κανονισμό του 2016 του 2008 στην πράξη η Ένωση ήδη εξασφάλισε εσωτερική εναρμόνιση για τους κανόνες αυτούς. Δηλαδή έχουμε προετοιμάσει το έδαφος για τη συμφωνία αυτή Ένωσης Καναδά. Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν ήδη το 2004 και η συμφωνία αναφέρεται στην αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιήσεων σε θέματα πολιτικής αεροπορίας και σε συμβατότητα μέτρων για το περιβάλλον. Ο στόχος είναι να διευκολυνθεί το εμπόριο προϊόντων και υπηρεσιών και υπάρχουν δύο βασικές πτυχές διαστάσεις στην συμφωνία αυτή. Πρώτον να διευκολυνθούν οι η έγκριση έτσι ώστε προϊόντα που να μπορούν να ε, ορίζονται οι άλλα που επισκευές και λοιπά με βάση το ένα ή το άλλο σύστημα να γίνονται με βάση τις ρυθμιστικές αρχές που ισχύουν και στην άλλη πλευρά. Και το δεύτερο, δεύτερο, το δεύτερο στοιχείο αναφέρεται στη συντήρηση που μπορεί να γίνεται από οργανισμούς που υφίστανται τον έλεγχο της άλλης πλευράς. Η προτινόμενη συμφωνία δείχνει την ε, βούληση του Καναδά για αμοιβαία, πλήρη αμοιβαία αναγνώριση και αποδοχή σε θέματα συντήρησης. Υπάρχουν επίσης αντίστοιχοι μηχανισμοί για συνεργασία και διαβούλευση σε θέματα ελέγχων, κοινοποιήσεις κλπ. Ένα συνεχές σύστημα εποπτείας της συμφωνίας επίσης υπάρχει Ήδη ο Καναδάς ανέλαβε να κάνει μια ανάλυση της ε, ασφάλειας για εταιρείε που ρυθμίζονται από τον οργανισμό Transport Canada και ενδεχομένως να προτείνουν και ορισμένα μέτρα όπου αυτό χρειάζεται. Η συμφωνία μπορεί αργότερα να υποστεί αλλαγή με μια πλήρη διαδικασία. Μια ανταλλαγή ε, κειμένων διπλωματικής χρειάς εκ μέρους των δύο πλευρών. Ο στόχος, όπως υπόθηκε, είναι να μειωθεί και η γραφειοκρατία και πιστεύω ότι όλες αυτές οι αλλαγές θα κοινοποιούνται, υποθέτω, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό να ζητήσουμε από την Κομισιό να μας στηρεί ενήμερους οτιδήποτε αλλαγών. Η, η συμφωνία αυτή είναι πολύ φιλόδοξη και είναι και πολύ γενναιόδορη. δεν υπήρχαν παρόμοιοι όροι στη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην περίπτωση δε της Βραζιλίας και εκεί υπάρχουν ορισμένε διατάξεις που δεν είναι τόσο φιλόδοξες. Όσο έχει βέβαια η συμφωνία αυτή είναι ένα πρώτο σήμα, κατά κάποιο τρόπο, ένα πρώτο παράδειγμα υπό τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Αυτά και οι συνάδελφοι αν έχουν να κάνουν σχόλια, εδώ είμαστε. πρόεδρο. Ευχαριστούμε κυρία Τικάου και για την τεχνική δουλειά που κάνετε για ένα θέμα που όντω είναι μια πρεμιέρα και όντω θα είναι παράδειγμα. Ο συνάδελφο Γκρό ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το θέμα αυτό, ξέρω, γιατί πήρε μέρο στι διαπραγματεύσει με τι ΗΠΑ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την συγκίτρια και την Επιτροπή για αυτή την ενημέρωση. Ε, δεν θα ήθελα να αναφερθώ τώρα σε τεχνικέ ε, λεπτομέρειε σε αυτό το ζήτημα. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τα όσα αναφέρει στο, ανέφερε στο τέλο η, η συγκίτρια, δηλαδή με βάση την προφορική ενημέρωση που λάβαμε. Θα ήθελα να λάβουμε και κάτι γραπτό ούτω ώστε να μπορούσαμε να κάνουμε μια σωστή συζήτηση εδώ. Με βάση τις πληροφορικέ ε, πληροφορίες που λάβαμε, η συμφωνία αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει υπόδειγμα για άλλες ε, συμφωνίε που θα ακολουθήσουν. Και θα το πω όταν θα είναι εδώ και εκπρόσωπος τη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι δεν ε, επαρκεί απλά το να έχει δείξει μια καλή πρόθεση ο, ο εταίρος. Θα πρέπει δηλαδή πραγματικά να συναυθεί μια συμφωνία ώστε να μπορέσουμε να αναφερθούμε σε κάτι τέτοιο. Θα πρέπει ε, να δούμε ε, τι ακριβώς περιμένουμε και τι ακριβώς θεωρούμε εμείς ως μια καλή ποιότητα σε συμφωνία. Θα πρέπει να θέσουμε ερωτήματα πιο συγκεκριμένα σε σχέση με αυτή τη συμφωνία όταν σας λέω θα έχουμε λάβει και γραπτός πλέον το κείμενό της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Κύριε Μέστερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ πολύ σύντομα. Ότι συμφωνούμε πλήρως ε, με τον ε, Μάτιο Γκος ε, σε αυτό που είπε ότι θα μπορούσε να αποτελέσει υπόδειγμα αυτή τη συμφωνία και ειδικότερα και για την συμφωνία με, την, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα έπρεπε οι Ηνωμένες Πολιτείες να διαβάσουν για να παραδειγματιστούν. Ένα ακόμα το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό είναι αυτό που ανέφερε και ο Ματιό Κρός, δηλαδή το ζήτημα α, το, της ε, συντήρησης του μηχανού. Δηλαδή, φυσικά αναμένουμε να δούμε και το κείμενο γραπτά πλέον της ε, πρότασης, αλλά πραγματικά αυτό το ζήτημα είναι πολύ σημαντικό ε, και όσο αφορά, όσον αφορά και τη θέσπιση σχετικών προτύπων για τις συντήρηση, των μηχανών, γιατί πραγματικά είναι πολύ ε, σημαντικό για ζητήματα ασφαλείας. Ε, άρα λοιπόν αναμένουμε και εμείς με ενδιαφέρον το τι ακριβώς θα αναφέρεται στο κείμενο και ευχαριστούμε βέβαια και την κυρία Τικάου για όλο το ενδιαφέρον που έχει δείξει. Ευχαριστώ κύριε Ευχαριστώ. Θα ήθελα να θέσω κάποια ερωτήματα από την πλευρά μου στην ε, Επιτροπή, καταρχήν σε ό,τι αφορά την αμοιβαιότητα ε, στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας για την ε, ασφάλεια στον αέριο χώρο. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι έλεγχοι ασφαλείας που έγιναν στον Καναδά ή σε άλλες χώρες αεροπορικές εταιρείες, ευρωπαϊκές ή αεροσκάφη ε, είχαν ε, επιδείξει προβλήματα στο πλαίσιο δηλαδή τέτοιων ε, ελέγχων ασφαλείας στο πλαίσιο της συμφωνίας ΑΦΑ είχε προβλεφθεί ότι πράγματι θα υπάρχουν έλεγχοι στους οποίους θα υποβάλλονται και οι εταιρείε και τα αεροσκάφη της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε καλό θα ήταν να γνωρίζουμε αν έχει γίνει κάτι τέτοιο στο παρελθόν. Είναι σημαντικό για την αμοιβή αναγνώριση των προτύπων. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα. Ε, θίγουν ζητήματα ε, safety, εσωτερικής, α το πούμε έτσι, ασφάλειας, ε, αυτές τι συμφωνίες ή και εξωτερική ασφάλειας, security. Και τρίτο ερώτημα. στο πλαίσιο μιας συμφωνία, συμφωνίας ε, για την ασφάλεια. Ε, για παράδειγμα, θίγονται και ζητήματα χρόνων ανάπαυσης ε, των πληρωμάτων και των πιλότων, γιατί βέβαια αποτελεί και αυτό ένα πολύ σημαντικό ζήτημα των logistics σε αυτήν την περίπτωση και γνωρίζουμε ότι από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού εκεί τα πρότυπα που ακολουθούνται είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λίστερμπεργκερ και Πράτμο. Ευχαριστώ. Θα κάνω δύο ε, μόνο σχόλια. Ε, λίγο με αυτό που είπε ο κύριος ε, Γκρόσε για τα αμερικανικά αγγλικά. Ε, τα αγγλικά είναι αγγλικά, έτσι. Και νομίζω πως ε, οι Αμερικανοί μπορούν να καταλάβουν τα αγγλικά, τα δικά μας, ας το πούμε έτσι. Τώρα, ένα δύο ε, σχόλια που θα ήθελα να κάνω αφορούν περισσότερο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρά τα σχόλια που έκανε η συγκεκριά μας. Άκουσα με ενδιαφέρον ε, αυτό που μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η συμφωνία δηλαδή έχει συνδυαστεί με στόχο την μείωση του γραφειοκρατία. της γραφειοκρατίας. Α, ε, στο ε, παρελθόν ε, βέβαια όταν είχαμε ασχοληθεί και με το ζήτημα της ΕΑΣΑ είδαμε τελικά ότι το γραφειοκρατικό της εργασίας αυξήθηκε αντί να μειωθεί. επειδή τώρα εγώ ήμουν επικεφαλής τη μια Επιτροπής επιτροπή για τη συνεργασία με τον Καναδά, ήθελα να να αναφερθώ ε, στο ότι ήταν σημαντική αυτή η διαφοροποίηση που έκανε η εισηγήτρια ανάμεσα στη Συμφωνία για την Ασφάλεια από αφενός και στην ε, ε, Συμφωνία για τις Υπηρεσίες Αφετέρου και θα ήθελα να ακούσω πώς έχει σχεδιαστεί αυτή η συμφωνία ώστε να υπάρχει διάδραση, να υπάρχει συνεργασία, στο πούμε έτσι, σχέδιση με την ε, συμφωνία, με την εμπορική συμφωνία που ε, διαπραγματευόμαστε αυτή την περίοδο με τον Καναδά. Και όπως είπε ο κύριος Καλέα στο πλαίσιο τους, ε, του αυξανόμενου εμπορικού όγκου μεταξύ Καναδά και Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να υπάρχει συσχέτιση, να υπάρχει σχέση μεταξύ αυτών των επιμέρων συμφωνιών και με μια γενικότερη εμπορική συμφωνία που θα ακολουθήσει. Και όπως είπε επίσης ο κύριος Γαλέτια, θα πρέπει να εξετάσουμε αυτό το ζήτημα στο πλαίσιο της ευρύτερης προοπτική που έχουμε για τη Βόρεια Αμερική ε, και στο πλαίσιο της μονογραφικής της Συμφωνίας Ασφαλείας με, την, ε, με ΗΠΑ. Υπάρχουν εκεί κοινά, κοινά σύνορα και χερσαία και ένα αέρια μεταξύ Καναδά και Πολιτειών και κατά συνέπεια δεν μπορούμε να ε, αντιμετωπίσουμε ξεχωριστά αυτέ τι δύο συμφωνίε και αυτέ τι δύο χώρε. Θα πρέπει να ζούμε ω ένα συνολικό πακέτο. Άρα λοιπόν το δικό μου ερώτημα είναι πώ αυτέ οι συμφωνίε θα ευθυγραμμιστούν, αν θέλετε, με μία ενδεχόμενη ευρεία ε, συμφωνία εμπορικού χαρακτήρα. Και ε, θα ήθελα να με διαβεβαιώσει πράγματι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι όταν μα λέει ότι θα μειωθεί η γραφειοκρατία, πράγματι θα μειωθεί. Σα ευχαριστούμε. Να δώσουμε το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, έτσι ώστε να απαντήσει και σε ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με το παραδειγματικό χαρακτήρα της συμφωνίας αυτής και αν υπάρχει δυνατότητα να επηρεάσουμε θετικά τις ε, σημερινές συμφωνίες ε, για τις ε, πτυχές μείωσης της γραφειοκρατίας, ελέγχου και να σχολιάσετε και τη σχέση μεταξύ safety και security. θέλουμε να δούμε αν υπάρχει ενδιαφέρον να ακολουθήσουμε ένα τέτοιο μοντέλο και στο μέλλον. Thank you very much. And I... Ευχαριστώ πολύ. Θα ε, προσπαθήσω να απαντήσω στα διάφορα ερωτήματα που τέθηκαν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν την κυρία Ρατικάου γιατί εξήγησε με πολύ καλό τρόπο το πλαίσιο στο οποίο γίνεται αυτή η συζήτηση. Έχουμε αυτή τη συμφωνία για την ασφάλεια η οποία την οποία διαπραγματεύτηκε ε, με δική της αποκλειστική αρμοδιότητα Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και εδώ έχουμε το πλεονέκτημα ε, σε αντίθεση δηλαδή με τις συμφωνίες εκείνες που χρήζουν εθνικής επικύρωσης ότι μπορούμε να προχωρήσουμε γρηγορότερα εφόσον δώσει τη σύμφωνη γνώμη του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα απαντήσω θετικά στο αίτημα της κυρίας Μάσα και του κυρίου Γκρός δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα λάβει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Είναι αρκετά τεχνικέ διαπραγματεύσει οι οποίε γίνονται, για παράδειγμα τεχνικά ζητήματα σε ό,τι αφορά την πιστοποίηση, τη συντήρηση και ούτω καθεξή. Αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα, μπορούμε να σα διαβιβάσουμε όλε αυτέ τι ε, πληροφορίε και οι συνάδελφοί μου που είναι εμπειρογνώμονε σε αυτά τα ζητήματα θα σα ε, παράσχουν όποιε πληροφορίε χρειάζεστε. Δεν υπάρχει πρόβλημα εδώ. Η κυρία Λίχτεμπεργκερ ε, έθεσε ένα ερώτημα σε ό,τι αφορά την αμοιβαιότητα στο πλαίσιο αυτή τη συμφωνία. Είναι πολύ σημαντική αυτή η πτυχή και θέλω να την ευχαριστήσω που την έδειξε. Γιατί ο στόχο μα στο πλαίσιο αυτή τη συμφωνία είναι ακριβώ αυτό. Η αμοιβαία αναγνώριση τη επιστοποίηση των προϊόντων. Αυτό δηλαδή που θα πρέπει να θυμόσαστε είναι ότι η συμφωνία αυτή προβλέπει την αμοιβαία αναγνώριση των επιστοποιήσεων, των πορισμάτων και των εγκρίσεων σε ό,τι αφορά την δυνατότητα ενός αεροσκάφους να, να λειτουργεί, το ζήτημα της καλής λειτουργίας, ε, συντήρησης, ε, ασφάλειας ε, των προϊόντων της αεροναφυγικής. Άρα λοιπόν αυτό στο οποίο συμφωνούμε με τον Καναδά είναι ότι θα υπάρχουν συμβατές μεταξύ τους διαδικασίες σε ό,τι αφορά τις τεχνικές προϋποθέσεις. Εφόσον αυτές οι τεχνικές προϋποθέσεις θα ισχύουν, θα είναι δυνατόν να επικυρώνονται αμοιβαία συγκεκριμένε πιστοποιήσει, πράγμα που είναι προ όφελό μα γιατί δεν χρειάζεται να πιστοποιούμε από εκεί και μετά ξανά και ξανά ήδη πιστοποιημένα προϊόντα, πρότυπα και ούτω καθεξή. Αυτό λοιπόν είναι προ όφελο και, και, και του κλάδου, γιατί δεν θα χρειάζεται να κάθε ξεχωριστό προϊόν να διέρχεται ξανά τη διαδικασία της επαναπιστοποίησης, ας το πούμε έτσι. Η κυρία να μας ρώτησε τώρα κατά πόσο θα είμαστε σίγουροι ότι αυτά τα πρότυπα θα είναι πράγματι σύμβατα μεταξύ τους, θα είναι συγκρίσιμα. Στη διαφορετική περίπτωση θα βάλουμε σε κίνδυνο την ασφάλειά μας. Να πω ότι λοιπόν έχουμε εμείς εντατικές συζητήσει με του εμπειρογνώμους, με την καναδική ε, πλευρά και είναι σημαντικό να πούμε ότι είδαμε μεγαλύτερες ομοιότητες εδώ μεταξύ δηλαδή των δικών μας κανόνων ασφαλείας σε σύγκριση με τις ομοιότητες που βρήκαμε σε σχέση με τις ε, Ηνωμένε Πολιτείε. Μιλάμε εδώ για κάποιους πολύ βασικούς εταίρους. Έτσι. Μιλάμε για τις Ηνωμένε Πολιτείε, τον Καναδά, τη Βραζιλία. Δεν θα δείτε δηλαδή ε, σωρία τέτοιων συμφωνιών τις οποίες σας ε, προτείνουμε. Προτού λοιπόν προτούμε, να προβούμε στη σύναψη άλλων αντίστοιχων συμφωνιών, θα πρέπει να κάνουμε αυτό που είπε σωστά κυρία Λίχτινμπεργκερ, δηλαδή ότι τα συγκεκριμένα πρότυπα ασφαλεία θα είναι συγκρίσιμα. Και αυτό έγινε στο πλαίσιο διαβουλεύσεων μεταξύ εμπειρογνωμόνων, αλλά όχι μόνο αυτό κάναμε, αλλά προκειμένου να αυξηθεί η αξιοπιστία στα συστήματα τη ε, κάθε πλευρά, ε, προβλέπονται αμοιβαίοι έλεγχοι και εμπιστεύσει ε, των ε, δεδομένων και από τις δύο πλευρές συμπεριλαμβανομένων και πληροφοριών σε ό,τι αφορά ατυχήματα και δεν υπάρχουν προβλήματα. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Ε, ε, αντίθετα υπάρχει ενδιαφέρον και από τους, από τους αρμόδιους και από τον κλάδο για την ανταλλαγή των πληροφοριών και πραγματικά δεν υπάρχει πρόβλημα και από την πλευρά του Καναδά. Επίση, να πω πως γίνονται διαβουλεύσει σε τεχνικό επίπεδο για την επίλυση προβλημάτων ή ζητημάτων προτού καταστούν προβλήματα. Δηλαδή εφόσον διακρίνουμε ότι υπάρχει κάποια διαφοροποίηση στι ε, στις μα μας ε, εργαζόμαστε επ' αυτόν και υπάρχει, υπάρχουν επιτροπές και υποεπιτροπές που εργάζονται επί συγκεκριμένων ζητημάτων του παρατήματος, ε, ε, ιδιαίτερα ε, τεχνικού χαρακτήρα για ζητήματα πιστοποίησης που θα μας επιτρέψουν να προχωρήσουμε προς τα εμπρός. Εάν υπάρξει κάποιο σημείο όπου υπάρχουν αμφιβολίες μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τα όσα προβλέπονται στη συμφωνία και από εκεί και μετά υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί που μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε την κατάσταση. Η κυρία Λίχτεμπεργκερ έθεσε επίσης το ερώτημα άλλων παραγόντων που μπορούν να έχουν εδώ μια επίπτωση. Για παράδειγμα, χρόνια ανάπαυση ε, πιλότων. Όχι, δεν περιλαμβάνονται στην ελόγω συμφωνία, γιατί μιλάμε για συμφωνία αναγνώριση πιστοποίησεων, αλλά μπορούμε από εκεί και μετά να την διευρύνουμε και σε άλλου ε, τομεί και αυτό προβλέπεται, δηλαδή τέτοια δυνατότητα διεύρυνση, επέκταση σε άλλου τομεί τη ε, συμφωνία μέσω ε, ε, επιπρόσθετων παρατημάτων, εφόσον το επιθυμούν και οι Καναδοί, αλλά υπάρχει ενδιαφέρον από την καναδική πλευρά, γιατί προφανώ πρόκειται για ένα ζήτημα σημαντικό για τα πληρώματα και για του επιλότου. Επίση αναφερθήκατε στο ζήτημα του security, τη ασφάλειας από εξωτερικού, ε, Όχι, δεν καλύπτεται από αυτή τη συμφωνία. Εδώ καλύπτεται μόνο το safety Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ στα ζητήματα που έθεσε ο κύριος Μπράντμπορν. Καταρχήν έθεσε ένα πρώτο ερώτημα. Είμαστε σίγουροι, μας ερώτησε ότι αυτή η συμφωνία θα μειώσει το γραφειοκρατικό φόρτο εργασίας. Ναι, απαντούμε, γιατί θα έχουμε τη δυνατότητα να ε, επαληθεύσουμε, να επικυρώσουμε τις ε, διαδικασίες ε, της άλλης πλευράς. Ήδη η δημιουργία της ΕΑΣΑ συνεπάγεται την ε, μείωση, την μεγάλη μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου εργασία στο πλαίσιο των πιστοποιήσεων. Ε, προ, προ, προ, προτού δημιουργηθεί αυτή η υπηρεσία, είχαμε ένα σύστημα αμοιβαία πιστοποίηση όπου έπρεπε κανεί να απευθυνθεί σε εθνικέ αρμόδιε αρχέ, που σημαίνει έπρεπε να απευθυνθεί σε 27 διαφορετικέ αρμόδιε αρχέ. Αλλά τώρα τι γίνεται. Πηγαίνει κανεί σε αυτή την υπηρεσία και μόνο σε αυτήν, πράγμα το οποίο σημαίνει βέβαια μείωση του σχετικού κόστους, μείωση του σχετικού φόρτου εργασίας. Και αν ρωτήσετε τον ε, κλάδο, θα σας πει, πέρα από κάποιες μικρέ επιχειρήσεις που πράγματι δεν το αρνούν, έχουν κάποια προβλήματα, αποτελεί λοιπόν μεγάλη βελτίωση και έχουμε μέσω αυτής της αυξημένης ασφάλειας και λιγότερη γραφειοκρατία. Αλλά με αυτή τη συμφωνία με τον Καναδά θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη μείωση της γραφειοκρατίας γιατί δεν θα χρειάζεται καν να πιστοποιούμε τα προϊόντα της καναδικής πλευράς για δεύτερη φορά. Θα υπάρχει αμοιβαία επικύρωση, αμοιβαία και για τα δικά μας προϊόντα τα οποία εξάγουμε προς τον Καναδά. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική. σημαντικό αυτό το επίτευγμα και είναι σημαντικό το οικονομικό όφελος. Τώρα, ποια η σχέση μεταξύ της, ε, της ε, παρούσας συμφωνίας ε, και των διαπραγματεύσεων για μια οικονομική και πολιτική συμφωνία. Ο, σωστά έδειξε ο κύριος Έμπραντμον. Ναι, θα πρέπει να ληφθεί αυτή η παράμετρος υπόψη, αλλά εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο της συνεργασίας. Έχουμε μια νομική βάση για τις μεταφορές, αφορούν δηλαδή συγκεκριμένα αυτό το βλάδο, ε, και αυτή είναι η νομική βάση την οποία χρησιμοποιούμε. Ε, ο νομέα, δηλαδή τη ενέργεια κυκλοφορία γενικά δεν ε, συμπεριλαμβάνεται και στου ε, τομεί του ΠΟΕ. Είναι κάτι το διαφορετικό. Αλλά αποτελεί ένα πολύ σημαντικό τμήμα του εμπορικού όγκου μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Καναδά, αφού αποτελούν δύο από του μεγαλύτερου κατασκευαστέ Άρα λοιπόν, ναι, στο πλαίσιο των ε, δραστηριοτήτων κορυφών που γίνονται σε ό,τι αφορά μια μελλοντική οικονομική και πολιτική συμφωνία, θίγονται αυτέ οι επιμέρου συμφωνίε. Και αναφέρεται ότι υπάρχουν και ωφέλη σε ό,τι αφορά και τη δημιουργία θέσεων εργασία. Και το καταξή. Ε, τώρα, το κατά πόσο θα μπορούσαμε να εντάξουμε μια τέτοια συμφωνία στο πλαίσιο μια ευρύτερη συμφωνία αμπρέλα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δούμε. Ε, προς το παρόν παραμένουν συμπληρωματικέ. Τέτοιε ε, συμφωνίες όπως η παρούσα ε, προς μια συμφωνία οικονομική και εμπορική. Εάν καταφέρουμε, αφού ε, απελευθερωθεί πλήρω ο, ο κλάδος αυτός και έχουμε τη δυνατότητα να προβλήσουμε στις σχετικέ επενδύσει. τότε θα πρέπει να κάνουμε αυτό που είπε ο κ. Μπράντμπορν, δηλαδή θα πρέπει τι συμφωνίε να συμπεριληφθούν σε μια ευρύτερη οικονομικού χαρακτήρα συμφωνία. Ένα τελευταίο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω αφορά την ε, συμφωνία για την ασφάλεια μεταξύ Ένωση και ΗΠΑ. Γνωρίζετε πω ήταν η πρώτη συμφωνία την οποία είχαμε διαπραγματευτεί αλλά δεν θα επικυρωθεί και δεν θα διαβιβαστεί για ακύρωση από τα κράτη-μέλη εάν δεν επιληθεί το ζήτημα των σταθμών επισκευής ε, στην Αυλαπή Foreign Repair Stations. Ε, δηλαδή, ακούσαμε πως ε, στο κογκρέσο προχωράνε τα πράγματα, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Προ το παρόν η συμφωνία πάντως αυτή μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο γιατί προχωράμε με την καναδική πλευρά και Ε, μπορεί να έχει θετικέ επιπτώσει γιατί και ο κλάδο από την πλευρά τη ε, Ευρώπη και της, ε, των Πολιτειών θέλει να προχωρήσουν τα πράγματα. Και είπε σωστά ο κύριο Ζεμπράτμπορν ότι όταν μιλάμε για την ευρωπαϊκή αγορά, μιλάμε για μια νέα αγορά. Οπότε θα πρέπει να συζητήσουμε και με, τις, με τις και με τον Καναδά αν θα μπορούσαμε να έχουμε μια συνολικότερη αν θέλετε, προσέγγιση με το Βόρειο Ατλαντικό. Αλλά ε, καταρχήν θα πρέπει να επιλύσουμε αυτό το ζήτημα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και βέβαια να δούμε και τι θα γίνει με τη Βραζιλία γιατί αποτελεί και αυτή μια μεγάλη προτεραιότητα. Ευχαριστώ πολύ. Και κάτι για να κλείσουμε. Είσαι κίτρια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους τοποθετήθηκαν ε, σήμερα και τους εκπροσώπους της Κομισιόν για τις απαντήσεις. Θα ήθελα να πω ότι το άρθρο 6 της συμφωνίας κάνει λόγο για safeguarding measures, μέτρα διασφάλισης και αναφέρεται σε προβληματικές καταστάσεις, δηλαδή στα προβλήματα που έχουμε με ορισμένες πιστοποίησεις που δίνονται από κάποιες αρχές έτσι ώστε όλοι να μπορούν να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα. Έχουμε λοιπόν αυτές τις ε, ρήτρες διασφάλισης. Και θα ήθελα να σας παραπέμψω και στο άρθρο 4, το οποίο καθορίζει το πεδίο εφαρμογής τη συμφωνίας. Η συμφωνία αυτή εφαρμόζεται στην εποπτεία της ε, πολιτικής αρχής ε, στην ε, έγκριση των καταστάσεων συντήρησης, των μονάδων συντήρησης, των μονάδων, των περιβαλλοντικών μονάδων και περιβαλλοντικής πιστοποίησης. Και έτσι λοιπόν θα πρέπει να το δούμε σε στενή σχέση με τη Συμφωνία Πλαίσιο για τους κοινούς κανόνες ε, για την, αστική, για την πολιτική αεροπορία. Και μπορούμε να λάβουμε και ορισμένα μέτρα που αναφέρθηκαν από την κυρία Λιχτεμπέργκερ. Θα ήθελα να σας, να σας ευχαριστήσω όλους για τις απόψεις σας και θα σας αναφέρω και κάποιες ημερομηνίες. Η έκθεση θα στέλνει για μετάφραση στις 3 Σεπτεμβρίου. Στις 27 Σεπτεμβρίου θα συζητήσουμε την έκθεση στην Επιτροπή μας και στη συνέχεια θα έχουμε τροπολογ... την κατάθεση τροπολογιών μέχρι τις 5 Οκτωβρίου. Θα υιοθετηθεί η έκθεση στην Επιτροπή στις 26 Οκτωβρίου και κάποια στιγμή στην Ολομελία του Νοεμβρίου, μάλλον στις 22. Ελπίζω να μπορέσω να τηρήσω αυτό το χρονοδιάγραμμα, καθώς ε, η πρόθεσή μας είναι να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ευχαριστούμε την κυρία Τικάου. Τα σημειώσαμε όλα αυτά. Σημειώσαμε και το ότι θα συζητηθεί στις 27 Σεπτεμβρίου η έκθεση και η ημερομηνία για την κατάθεση τροπολογιών είναι 5η Οκτωβρίου. Ας περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο της για να ολοκληρώσουμε την πρωινή μα συνεδρίαση. Λογικά μας φτάνει ο χρόνος. Ξέρετε ότι τα ευρωπαϊκά δίκτυα, ευρωπαϊκά εγγράφονται σε ενα πολυετες πολιετές ε, σχέδιο 2007-2008. Αυτά τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενδιαφέρουν ε, όλους τους τρόπους μεταφοράς και σε ό,τι αφορά τώρα την διαχείριση της ενέργειας κυκλοφορίας έχουμε το σύστημα ATM, το σύστημα το, το οποίο διαχειρίζεται λειτουργικά τμήματα του ενεργείου χώρου που πρέπει να μεταρρυθμιστούν αυτά τα FABs, ε, όπως λέγονται, αυτά τα λειτουργικά μπλοκ εμπίπτουν στην επιτροπολογία και έχει και το Κοινοβούλιο δικαίωμα ε, εξέτασης ε, όμως ε, έγινε παραδεκτό ότι η Κομισιόν θα έρχονταν εδώ να μας κοινοποιήσει τους διαγωνισμούς που προκυρήσει για αυτά τα λειτουργικά τμήματα. Το 2010 είχαμε αξία για 20 εκατομμύρια ευρώ θα παρουσιαστεί από την Κομισιόν. Έρθουν εδώ ο αρμόδιο της Κομισιόν, ο αρμόδιο εκπροσωπικό Κομισιόν, ο κύριο Πακέ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να παρουσιάσω τα αποτελέσματα της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τα λειτουργικά τμήματα του εναερίου χώρου στα πλαίσια του πολιετούς προγράμματος για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών που ε, ξεκίνησε το 2010. Συμφων... Είχε γίνει μια συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής για τον Προπολογισμό και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η συμφωνία ήταν ότι η Κομισιόν θα παρουσίασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα αποτελέσματα των ε, προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και την επιλογή των έργων που σκόπευε να υιοθετήσει η Κομισιόν πριν να έχουν υποβληθεί αυτά στα ε, κράτη-μέλη και πριν να ξεκινήσει η επίσημη διαδικασία του δικαιώματο εξέταση. Έτσι λοιπόν σας παρουσιάζουμε τώρα αυτά τα πρώτα αποτελέσματα των διαγωνισμών 2010 ε, πριν από τις 15 ε, Ιουλίου να τα παρουσιάσουμε στα κρατη μπελη Τώρα οι διαγωνισμοί για το 2010 είναι τρεις. Έχουμε το πολιτες πρόγραμμα με μια συνιστός ATM Fabs που συζητούμε σήμερα αλλά και με δύο συνιστώσεις ε, αυτοκινητόδρομοι της ε, θάλασσας και ε, υπηρεσίες ενημέρωσης για τις πλωτές μεταφορές. Έχουν ξεκινήσει οι διαγωνισμοί και τα project θα υποβληθούν στις 30 Αυγούστου, ενώ η διαδικασία επιλογής θα λάβει χώρα το φθινόπωρο και θα επανέλθουμε προς το Ευρωπαϊκό, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα κράτη-μέλη περί τα τέλη Νοεμβρίου για τα αποτελέσματα. Τώρα η δεύτερη πρόσκληση υποβολή προτάσεων ε, που τρέχει αφορά το, ε, το πρόγραμμα που ε, τρέχει κάθε έτος και φέτος καλύπτει διάφορες πτυχές. Το πρόγραμμα εργασίας εξετάστηκε από αυτή την Επιτροπή και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καλύπτει αφενός μέτρα που έχουν να κάνουν με τις ΔΙΤ και επίσης ε, καλύπτει μελέτες που θέλουν να ευνοήσουν την ανάδυση ε, έργων κοινού ενδιαφέροντος για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και επίσης στοχεύουν στο να ευνοήσουν κάποια γενοτόμα μέτρα προκειμένου να προωθήσουμε την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφορών κυρίως υπό τη μορφή μέτρων που θα μπορούσαν ε, να προωθήσουν διατροπικές πλατφόρμες ή τεχνολογικής φύσεως μέτρα πιο καινοτόμα. Αυτό για το ετήσιο πρόγραμμα, το οποίο επίσης ε, ε, ε ουσιαστικά τρέχει, είναι ανοιχτός ο διαγωνισμός, ε, θα γίνει μια αξιολόγηση στο φθινόπωρο και θα επανέλθουμε όπως και για τις δύο άλλες πτυχές του πολιτούς προγράμματος περί τα τέλη Νοεμβρίου. Επίσης προωθήσαμε την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τα λειτουργικά τμήματα του ενέργειου χώρου ήδη τον Απρίλιο καθώς αυτό το σημαντικό project του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ουρανού ήταν πιο όριμο από τα υπόλοιπα και είχε κατατεθεί έτοιμα χρηματοδότηση στην Κομισιόν. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να αποσυνδέσουμε αυτό το διαγωνισμό από τους άλλους. Άνοιξε τον Απριλίο, η εξολόγηση έγινε Μάιο και Ιούνιο και τώρα μπορούμε να σας παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διανέμει μια μπροσούρα, ένα φυλάδιο. Νομίζω ότι τα έχουν τα μέλη τη Επιτροπή σας. Στο έγγραφο αυτό περιγράφεται η διαδικασία της αξιολόγηση. Ως συνήθως έχουμε εξωτερική αξιολόγηση από τους εμπειρογνώμονες που επέλεξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατόπιν έχουμε εσωτερικό πάνελ το οποίο καθορίζει τη διαδικασία της επιλογής που σας παρουσιάζεται σήμερα. Έχουμε διαθέσιμα 20 εκατομμύρια ευρώ, έχουμε 6 προτάσεις για ένα ποσό 35 εκατομμύριων ευρώ. Όπως, ε, ξέρετε, όπως βλέπετε ξεπεράστηκε ο προπολογισμό ό,τι αφορά τις εργασίες της εξωτερικής αξιολόγησης μας ε, έμεναν τέσσερα project, απορρίφθηκαν δύο και το ιστορικό πάνελ της Κομισιόν εξέτασε εκ νέων αυτά τα project και έτσι λοιπόν ε, ε, ουσιαστικά μειώσαμε το φάσμα, διατηρήσαμε τις δραστηριότητε για το 2011 και 2012, έτσι λοιπόν σεβαστήκαμε τον αρχικό προϋπολογισμό των 20 εκατομμυρίων. Η πρόταση λοιπόν που σοσιάζεται σήμερα αφορά τέσσερα project, τέσσερις αποφάσεις χρηματοδότησης, των οποίων ο στόχος είναι να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη αυτών των λειτουργικών τμήματων του ενέργου χώρου για το ΦΑΜΠΕΚ που είναι το πιο σημαντικό για 13 εκατομμύρια συνεισφορά για το ΦΑΜΠ UK Island ένα ε, εκατομμύριο ευρώ πρόταση χρηματοδότηση για το North European Functional Space Block, την FAB, και τελευταία πρόταση για το FAB της Κεντρικής Ευρώπης για 1,4 εκατομμύρια. Αυτές οι τέσσερις προτάσεις λοιπόν παρουσιάζονται σε σας προς έγκριση. Φτάνουμε στα 20,4 εκατομμύρια, δηλαδή λίγο παραπάνω από το αρχικό ενδεικτικό ποσό, αλλά το λέτε, προγράμματα φτάνουν στα 115 εκατομμύρια. Έτσι λοιπόν ε, έχουμε κάτι παραπάνω. Ε, αυτά τις 400.000 όμως δεν υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έτσι λοιπόν το έγγραφο αυτό θα συζητηθεί στη συνέχεια και με τα κρατημέλη και ελπίσουμε ότι κατόπιν της έγκρισης ε, που θα έχουμε από την Μουσιονομική Επιτροπή αυτή την Πέμπτη θα έχουμε και υιοθέτηση από την Κομισιόν το Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτεμβρίου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Πακέ. Αρχίζουμε με τον κύριο Γκρός. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτή την ενημέρωση. Ε, θα ήθελα να λάβω περισσότερες πληροφορίες σε ό,τι αφορά το πρώτο project, τα κριτήρια επιλογής. Έχουμε κάποιες πληροφορίες τις οποίες λάβαμε από αλλού και τις διαβάσαμε. Αλλά πέρα από το μοτοδοτικό πλαίσιο και τις συγκεκριμένες ε, προτάσεις που έγιναν από αυτή την πτυχή, δηλαδή την οικονομική, θα ήθελα να ξέρω ποια ήταν ακριβώς ε, τα κριτήρια ε, με βάση τα οποία έγινε η επιλογή και ποιοι είναι ακριβώς οι στόχοι των project, γιατί πραγματικά από τις πληροφορίες τις οποίες λάβαμε αυτά δεν είναι δυνατό να τα διαπιστώσουμε. Άρα λοιπόν θα θέλαμε, δηλαδή πέρα από το οικονομικό χρηματοδοτικό πλαίσιο, να δούμε εδώ και λίγα πράγματα επί του περιεχομένου για να μπορέσουμε να έχουμε μια άποψη ολοκληρωμένη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Γκρός. Ευχαριστώ πολύ. Στο ίδιο μήκο κύματο και εγώ θα ήθελα μερικέ λεπτομέρειε από την Κομισιόν για τα διάφορα επιμέρους προγράμματα προς επιδότηση. Δώστε μας περισσότερες πληροφορίες. Τι ακριβώς θα κάνουν τα FAB με τα χρήματα που θα πάρουν. Αυτό ήταν γίνει η ερώτηση. Μια δεύτερη ερώτηση τώρα. Τι ποσά ήδη δόθηκαν στα διάφορα μπλοκ τμήματα του ενέργειου χώρου. Αν έχει γίνει αυτό, έχει γίνει ήδη ή όχι. Και για τα επόμενα έτη τι προβλέπετε προκειμένου να λειτουργούν τα ε, τμήματα αυτά του ενέργειου χώρου. Και μια άλλη και αυτή γενική ερώτηση. Διαπιστώνω ότι υπάρχει ένα λειτουργικό τμήμα ενέργειου χώρου για το κέντρο της Ευρώπης. και αυτό το FAB θα, έχει, θα πάρει σημαντικά κονδύλια. Αυτό σημαίνει ότι αυτό βρίσκεται πιο μπροστά, έχει προχωρήσει περισσότερο από τα άλλα FAB. Και με τα άλλα FAB, λειτουργικά τμήματα, τι γίνεται. Τι σχέση δηλαδή υπάρχει στον βαθμό εξέλιξης και προώθησης των διαφόρων λειτουργικών τμήματων. Και θα ήθελα να να μας πείτε αν αυτό συμφωνεί με αυτό που είχατε προβλέψει στην αρχή. Και η κυρία Γιάννησεν. Στα αγγλικά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για αυτό το πολύ ενδιαφέρον υλικό. Προσυπογράφω και εγώ τις ερωτήσεις που έκαναν οι δύο προηγούμενοι συνάδελφοι και ευρύνω λίγο τη συζήτηση Το 2012 η προθεσμία αυτή θα τηρηθεί γιατί βλέποντας κανείς την εικόνα διαρωτάτε πού προχωράμε και πού δεν προχωράμε. Μπορείτε να μας κάνετε μια σύντομη επισκόπηση του πού τα πράγματα κινούνται πιο γρήγορα και πού φαίνεται να υπάρχουν προβλήματα. Και ένα σχόλιο. Για μια φορά ακόμη βλέπουμε ένα σωρό ιδέες για προγράμματα για τις μεταφορές, αλλά δεν υπάρχουν αρκετά λεφτά. Και πρέπει να είστε πολύ αυστηροί για τα 20 εκατομμύρια, που 20, ίσως να μην είναι καν 20 εκατομμύρια. Αυτό μας δείχνει όταν μιλάμε για τις δημοσιονομικές προοπτικές. Εδώ υπάρχει ένα συγκεκριμένο παράδειγμα ότι έχουμε δίκιο και μπορούμε να πούμε ότι έχουμε περισσότερα σοβαρά προγράμματα αλλά λιγότερα χρήματα σε σχέση με τα προγράμματα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Η κυρία Λίχτενμπεργκερ. Ja, herzlichen Dank. Ähm, auch für mich bleiben einige wesentliche. Και εγώ διαβάζοντας αυτό το κείμενο ε, έχω ακόμα κάποια ερωτήματα. Γιατί ε, σε κάποιους ε, τομείς ε, δεν διευκρινίζεται προς τα πού ακριβώς κατευθύνονται αυτά τα κονδύλια, σε τι χρησιμοποιούνται. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το σημείο ένα στο οποίο έρευσαν, να το πούμε έτσι, τα, το μεγαλύτερο τμήμα των κονδυλίων, δεν ε, καθίσταται σαφές το τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι η πρόοδος που επιτυγχάνεται σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση. Σε ό,τι αφορά το παγέτο 3, και αυτό το βόρειο ευρωπαϊκό μπλοκ ότι το activity ε, ε, package ε, system δεν επεκτείνεται σε ένα συγκεκριμένο τομέα γιατί δεν αποτελεί προτεραιότητα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς εννοείται. Μετά το μπλοκ 4, Κεντρική Ευρώπη, αντιλαμβάνομαι ότι πρόκειται για ένα περίπλοκο τομέα, γιατί εδώ ο εθνικισμός εντό εισαγωγικών έρχεται να δημιουργήσει κάποια προβλήματα, θεωρώ πως θα φτάσουμε σε μια λύση εδώ, σε μια καλή λύση, αλλά θα ήθελα να ξέρω γιατί η Σλοβακία δεν περιλαμβάνεται πλέον και τι θα συμβεί. Γιατί πραγματικά, εάν δω το χάρτη, ε, χωρί τη Σλοβακία, με το κοινό ας πούμε, τη Σλοβακία στη μέση, ε, ε, θα είναι πραγματικά πολύ, μα πολύ περίεργο αυτό το ΦΑΠ και πολύ περίεργο αυτό ο τομέα. Και όταν λέτε μετά, το να, όταν προτείνονται κάποια ένα σενάριο με βάση τον τομέα αρμοδιότητα, area of responsibility, δεν αντιλαμβάνομαι τι ακριβώ εννοείται και θα ήθελα να μου το εξηγήσετε. Εγώ αυτό που κατάλαβα είναι μια ενισχυμένη συνεργασία που θα ισχύσει. Δεν αντιλαμβάνομαι λοιπόν γιατί για μια τέτοια ενισχυμένη συνεργασία θα πρέπει να υπάρξει μια επιπρόσθετη χρηματοδότηση ταξης 1,5 ε, εκατομμυρίου ευρώ. Και έχω την αίσθηση ότι κινούμαστε λίγο αργά εδώ. Νομίζω πως ε, κάποια στιγμή θα πρέπει να δώσουμε μια προειδοποίηση να πούμε για παράδειγμα πείτε μας ότι δεν θέλετε να το κάνετε, ανακοινώστε το και αναλάβετε τις ευθύνες σας. Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Εδώ και χρόνια δηλαδή να λαμβάνουμε κάποιες εκθέσεις όπου δεν βλέπουμε να σημαίνονται πρόοδος και ο καθένας να προσπαθεί δηλαδή ε, να προωθήσει και να αναδείξει το δικό του φάπο στο καλύτερο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό για πάντα. και δεν θα μπορούσαμε να δεχτούμε, για παράδειγμα, την κύρια αρμοδιότητα ή έδρα για, τον έλεγχο του αέριου χώρου μιας ε, χώρας να βρίσκεται σε μια άλλη. Δεν θέλω να επιστρέψω σε περισσότερε λεπτομέρειε σε αυτό το ζήτημα. Πρόκειται για το πολυεθνικό θέμα, αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι δύσκολη. Είναι μια βραδιά διαδικασία, δεν βλέπουμε να σημειώνονται μεγάλες πρόοδοι και ερωτώ σε ποιους εναέρους ε, χώρους έχουμε και ε, τους ενόπλες δυνάμεις που εδώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Φώστερ. Yeah, thank you, Chairman, and thank you to the Commission for... Uh, Ευχαριστώ και ευχαριστώ και την ε, Κομισιόν που τοποθετήθηκε σήμερα για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Πριν λίγου μήνε, ε, ο Πατρική έκανε μια πολύ καλή παρουσίαση στην Επιτροπή και μα βοήθησε πολύ. Νομίζω όμω ότι γενικά υπάρχει μια σύγχυση <laughs> των περισσότερων και μάλλον ε, και εσεί είστε κάπω σύγχυσμένοι γιατί έχουμε καταναλώσει πολύ χρόνο. Ξεκίνησε με τον ενιαίο ουρανού και προχωρήσαμε στο ΣΕΣΑΡ. Όμως ε, δεν ε, κατανοούμε πολύ καλά τι ρόλο διαδραματίζει η βιομηχανία σε όλο αυτό. Ο κλάδος μάλλον. Έχω πάντως κάποιες ερωτήσεις. Ε, ποιο είπε η κυρία Λίχτεμπερκ ότι υπάρχουν καθυστερήσεις. Καταρχήν έχουμε το θέμα της χρηματοδότησης και θα έρθω σε αυτό. Όμως έχουμε και το θέμα των χωρών που εμπλέκονται σε κάθε συγκεκριμένο Δηλαδή για το ποιο πιέζει και προχωρά πέρα από το ότι πρέπει να υπάρχουν περισσότερες διευκρινήσεις ε, και να δούμε τελικά ποιος κάνει προσπάθεια και ποιος όχι γιατί αυτό δεν είναι αποδεκτό. Ξέρουμε ότι ορισμένε από τι περιοχέ FAB ε, εργάζονται σκληρά για να προχωρήσει όλο αυτό το project και το συζητήσαμε και την Ισπανική Προεδρία. Ένα από τα κύρια θέματα ήταν, με το οποίο ασχολήθηκαν ήταν όλο αυτό με την ηφαιστειακή τέφρα και προσπάθησαν ε, να ε, βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του ενέργειου χώρου και να μειωθεί το κόστος. Έτσι λοιπόν πρέπει να δούμε ποιος καθυστερεί. Σε ό,τι αφορά τώρα τη χρηματοδότηση αυτή καθ' αυτή, νομίζω ότι θυμάμαι ότι πριν κάποια χρόνια πέρα από τις οδούς χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαμε και ε, μία πρωτοβουλία που λεγόταν Clean Sky και εμπλέκονταν εκεί και οι φαρμακοβιομηχανίες και, υπήρχαν, ε, και υπήρχε εκεί συμμετοχή και από τον ιδιωτικό τομέα και από την Κομισιόν όμως υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη γραφειοκρατία ε, τρομερή γραφειοκρατία για τη χρηματοδότηση που ερχόταν από την ευρωπαϊκή πλευρά έτσι λοιπόν εδώ βέβαια εξετάζουμε την χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών δικτύων Βέβαια, μπορώ να καταλάβω το 0, 1, 2, 3. Κοιτάξτε, η Πολωνία είναι σχετικά νέο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι και μεγάλη χώρα. Δεν είναι πολύ ενθαρρυντικό να βλέπουμε ότι δεν κινείται τόσο γρήγορα όσο θα έπρεπε. Εδώ μιλάμε για οριμότητα. Όμως, ε, ε, εδώ που ανησυχώ, παραδείγματο χάρη, βλέπω πώς συμπεριφέρεται η Ιταλία. Δεν θέλω τώρα εδώ να δακτυλοδείξω τους Ιταλούς, αλλά σε αυτό το στάδιο του παιχνιδιού. Αναρωτιέμαι γιατί μια χώρα σαν την Ιταλία, μια προηγμένη χώρα, βρίσκεται τόσο χαμηλά στον κατάλογο. Η Ιταλία έχει κατασκευάσει πολύ καλά αεροσκάφη. Δεν χρειάζεται να την υπερασπίσω, αλλά απλώ εκπλήσωμαι που στην περίπτωση αυτή βλέπουμε αρνητικά αποτελέσματα. Γιατί η Ιταλία είναι πλήρε μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γιατί σε αυτή την κατηγορία εδώ κάνουν κάποιες δράσεις που δεν θα συστήνονταν. Τώρα, σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη χρηματοδότηση, αν δούμε τα διευρωπαϊκά δίκτυα, βλέπουμε την κατανομή με σαφήνεια. Όλα τα υπόλοιπα θα μπουν από τον κλάδο ή προέρχεται και κάποια χρηματοδότηση κατευθείαν από τα κράτη-μέλη. Γιατί ξέρουμε ότι έχουμε και τι εθνικέ υπηρεσίε, αλλά στον Ηνωμένο Βασίλειο έχει ιδιωτικοποιηθεί η υπηρεσία αυτή, παραδείγματο χάρη. Όμω ξέρουμε ότι σε ορισμένε χώρε ε, είναι δημόσιε υπηρεσίε. Είναι λοιπόν πολύ πλοκό το θέμα. Έτσι λοιπόν, αν μπορείτε να διευκρινίσετε αυτά τα σημεία, θα σας ευγνωμονούσα. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την κυρία Φώστερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ τον κύριο Πακή για την παρουσίασή του και επίσης να θέσω κάποιες ερωτήσεις. Θα ήθελα να ξέρω καταρχήν όπως φαίνεται από τα 8 μπλοκ, ε, μόνο οι έξι παρουσίασαν πρόταση. Θα ήθελα να πω γιατί παίρνουν το χάρη κάποιοι Πορτογαλία, Ισπανία ή το τμήμα του Δούναβη ή της Βαλτικής. Γιατί δεν παρουσίασαν ε, κάποιες προτάσεις. Μήπως μπορείτε να μας πείτε γιατί. Και από τους 6 ε, επιλέξατε τους 4, τα τέσσερα project. Ποιοι είναι οι λόγοι. Επειδή το Ιταλικό και το Πολωνικό αφορούσαν πολύ λίγα κράτη-μέλη. Ένα μόνο λόγω χάρη. Και σε ό,τι αφορά τα αριθμητικά στοιχεία. Στο πρώτο project, το οποίο λαμβάνει και τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση, Είχαμε 42% ποσοστό χρηματοδότηση ενώ αυτό που επιτυγχάνεται τελικά είναι σχεδόν το 50%. Εδώ θα ήθελα να μου πείτε γιατί από όλο το project έχουν τροποποιηθεί ουσιαστικά κάποια στοιχεία κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης. Λέγεται μάλιστα ότι ένα τμήμα άλλαξε κατηγορία και θεωρήθηκε ως ε, έργα δεν ξέρω τι σημαίνει ακριβώς αυτό. Τι εννοείται. Δηλαδή βλέπω δύο που είναι ένα μείγμα μεταξύ μελέτης και έργων ή εφαρμογής και άλλα που αφορούν μόνο μελέτες. Μήπως μπορείτε να μας το εξηγήσετε λίγο. Και μάλιστα επίσης βλέπουμε ότι κάποια από τα project ε, πάνε πέρα από το 2012. Αυτό ε, δεν αποτελεί των προηγούμενων ε, κριτηρίων γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις δεν χρησιμοποιήθηκε κάποιο τμήμα τη χρηματοδότηση. Και επίση για τη Σλοβακία αποφάσισε να μην συμμετάσχει στο διαγωνισμό και να μην συμμετάσχει στο project. Θα ήθελα να ξέρω για ποιο λόγο. Και επίση, να μας πείτε πότε θα μπορέσουμε να δούμε, να σημειώσουμε τις βελτιώσεις που θα έχουν γίνει σε σχέση με τα λειτουργικά τμήματα του εναέριου χώρου. Κύριε Κασίν. Ehm, Καταρχήν, θα ήθελα να συγχαρώ την Κομισιόν και για το διαγωνισμό που για τη, κατά τη γνώμη μου είναι μια καλή ευκαιρία για χώρες που, που είναι στα ΦΑΜ να απαντήσουν στο βασικό ερώτημα πώς θα γίνει η ενοποίηση μέσα σε αυτά τα λειτουργικά τμήματα. Τώρα μια συγκεκριμένη ερώτηση για τη λευκή ζώνη στα Βαλκάνια. Είναι το ανατολικό τμήμα της πρώην Ιουγκοσλαβίας. Σερβία, Μοντενέγκρο, Κόσοβο και Μακεδονία. Που δεν είναι τμήμα οποιοδήποτε, κανενός μάλλον από αυτά τα λειτουργικά τμήματα. Η συγγήτριά μας, είμαι εισηγητής για τη Σερβία και κάθε φορά που πάω στο Βελιγράδι συναντάω μια ομάδα ειδικών που βοηθάνε την κυβέρνηση εκεί στο να εναρμονίσει την νομοθεσία της και σε θέματα ε, ενέργειας κυκλοφορίας, ελέγχου ενέργειας κυκλοφορίας και θα ήθελα να μάθω αν σημειώθηκε κάποια πρόοδος, αν Είμαστε κοντά σε μια απόφαση που θα δίνει απάντηση στο ερώτημα θέλουν να έχουν δικό τους λειτουργικό τμήμα, δικό τους μπλοκ ή θέλουν να αποτελέσουν τμήμα του κεντρικού χώρου, κεντρικού τμήματος της Ευρώπης ή του τμήματος του Δουνάβεως. Μια δεύτερη πιο λειτουργική ερώτηση. Χαίρομαι για το ότι δύο μπλοκ ήδη συμπεριλαμβάνουν και την ε, δύο χώρες της Αφρικής, την Ίσια και Αίγυπτος αφενός, καλό αυτό, ιδιαίτερα όσον αφορά το μεσογειακό μπλε μπλοκ. Απ' την άλλη μεριά, για την Ισπανία, για την Πορτογαλία, βλέπουμε το Μαρόκο δεν συμπεριλαμβάνεται πουθενά. Και νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία να επεκτείνουμε το μπλοκ και για το Μαρόκο ιδιαίτερα λόγω της μεγάλης συχνότητας των πτήσεων και πάρα πολλοί τουρίστες πάνε στο Μαρόκο. Και τέλος, θυμίζω σε όλους μας ότι η Τουρκία είναι υποψήφια προς ένταξη χώρα και αν το μεσογειακό μπλοκ μπορούσε να συμπεριλάβει και την Τουρκία, γιατί όχι. Δεν θα ήταν κακό αυτό αυτό θα βοηθούσε την ασφάλεια στις αερομεταφορές. Παρακαλώ λοιπόν την Κομισιό να απαντήσει στο ερώτημά μου. Κυρίως, σκεφτήκατε να συμπεριλάβετε και κάποια άλλη χώρα σε οποιοδήποτε από τα μπλοκ που υπάρχουν και πιο συγκεκριμένα υποψήφιες προς ένταξη χώρες και ενδεχομένως χώρες που θα μπορούσαν να γίνουν υποψήφιες στο μέλλον. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Κύριε Ρόσμπαχ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τα όσα είπε ο κ. Κασίμ. Γιατί εγώ είμαι νέο μέλο αυτής τη Επιτροπής ε, και λόγω ενδεχομένω τη άγνοιά μου θα ρωτήσω αυτό που θα ρωτήσω. Οι περισσότερες από αυτές τις ε, χώρε που περιλαμβάνονται εδώ ούτε ευρωπαϊκέ ε, χώρε, ούτε υποψήφιες για ένταξη χώρε είναι. Ε, αναφέρομαι εδώ ειδικότερα στο βόρειο μπλοκ. Η Γρυλανδία έχει εξαιρεθεί, δεν δηλαδή θέλει να θεωρείται ευρωπαϊκό κράτο κράτος παρότι αποτελεί τμήμα της Δανίας. Άρα πώς θα γίνει ακριβώς η χρηματοδότηση. Μιλάμε δηλαδή για ένα μπλοκ εδώ που περιλαμβάνει την Ισλανδία, τη Γρυλανδία και την Ορβηγία, χώρες που δεν είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και δεν αντιλαμβάνω πώς θα γίνει η χρηματοδότηση σε αυτά τα μπλοκ. Ε, αλλά να πω κι εγώ ότι όπως ε, και, και άλλοι συνάδελφοι δεν έχουμε λάβει πολύ συγκεκριμένες ε, πληροφορίες ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα κριτήρια με τα οποία γίνεται η επιλογή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Τικάου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, εάν δούμε το ποσοστό συγχρηματοδότηση από τον προπολογισμό των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορά θα δούμε πω ε, ανέρχεται στο 50%. Άρα δηλαδή γιατί μιλάμε εδώ για κάποιες ε, μελέτες οι οποίες θα προσπαθήσουν να καθορίσουν τον, ε, το μέλλον των ε, φάψε, Αλλά δεν είδα πουθενά τίποτα για κατευθυντήρε γραμμές. Κατευθυντήρε γραμμές οι οποίες θα έπρεπε να είχαν εκπονηθεί σε ό,τι αφορά τον ορισμό αυτών καθεαυτών των FAP. Ε, θυμάμαι και σε σχέση με το σύστημα της Eurocontrol είχαμε θέσει το ίδιο ερώτημα και η απάντηση που είχαμε λάβει είναι ότι ως τα μέσα του 2010 θα έχουν οριστεί οι ειδικέ κατευθύντερες γραμμές. Πού είναι λοιπόν. Δεν τις έχω δει ακόμα. Ερωτώ λοιπόν, με βάση ποια κριτήρια θα οριστούν αυτά τα ΦΑΠ και πώ θα είναι δυνατόν να γίνει η χρηματοδότησή του χωρί να έχουν οριστεί τέτοια κριτήρια και κατευθύνσει γραμμέ. Σε ό,τι αφορά το FB του Δούναβε, θυμάμαι ότι στη σχετική απόφαση του 2009 είχε εγκριθεί η χρηματοδότηση για το Δούναβε και για άλλε περιοχέ. Και επειδή είχε εγκριθεί, είχαμε ζητήσει από την ε, Επιτροπή να μα ενημερώνει τακτικά ω προ τα όσα συμβαίνουν ε, και να μας ενημερώσει και ε, σε σχέση με τα πορίσματα των σχετικών ε, μελετών, εάν έχουν ολοκληρωθεί. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Μέσνερ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Με ενδιαφέρει αυτό το ζήτημα, ζήτημα γιατί δεν περιλαμβάνεται πλέον η Σλοβακία και όπω αναφέρθηκε από τον συνάδελφο, υπάρχουν και άλλε χώρε που δεν συμμετέχουν. Τι θα μπορούσαμε λοιπόν να κάνουμε να, για να συμπεριλάβουμε όλε αυτέ τι χώρε, γιατί αν μιλάμε για ευρωπαϊκό ένα αεροχώρο, τότε πραγματικά θα πρέπει να μιλάμε για όλε τι χώρε. Και μετά, ένα ακόμα ζήτημα που με απασχολεί και μια έλλειψη την οποία παρατήρησα είναι ε, μία ανάλυση σε ό,τι αφορά τις αδυναμίες ε, του ε, αέριου χώρου. Ε, δηλαδή αποτελεί μια καλή βάση το να έχουμε δει καταρχήν το τι λείπει, τι δεν λειτουργεί σωστά, τι μας χρειάζεται τόσο ώστε να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε. Κατάλληλα ίσως θα μπορέσει να μας πει κάτι ο πρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, παρατηρώντας ότι η συζήτηση έχει διευρυνθεί πολύ ε, και παρά το γεγονός ότι διστάζω θα θέσω δύο ερωτήματα που σε μια τόσο διευρυμένη συζήτηση για τα FABs μπορεί να φαίνονται ενδιαφέροντα. Ε, πρώτο θέμα, ε, θα ήθελα να γνωρίζω, διεκδικώντας ένα χρόνο από τις απαντήσεις της Επιτροπής, σε τι ακριβώς συνίσταται η συνεργασία πολιτικής και στρατιωτικής διάστασης στα FABs, πώς αυτή ε, υλοποιείται και ε, κατά πόσον οι ισχύοντες κανόνες στα πλαίσια του ICAO εφαρμόζονται μέχρι ποιο βαθμό και με ποιο συντονισμό ε, στα πλαίσια των ΦΑΒΣ. Ευχαριστώ πολύ. Euh, Ευχαριστούμε κύριε Κουμουτσάκο. Θα ξαναδώσουμε το λόγο στον κύριο Πακέ. Θα ήθελα να κάνω όμως και εγώ ένα σχόλιο. Είδαμε ότι έχουμε ένα σωρό ερωτήσει. Παρότι το θέμα είναι τεχνικό. Κάτι που παραξενεύει είναι το εξή. Εδώ έχουμε ένα χάρτη του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού. Περίεργο αυτό. Βέβαια υπάρχουν ιστορικά δεδομένα, τεχνικά δεδομένα για το κάθε ένα από αυτά τα μπλοκ. Αλλά και ο χάρτης, όταν μιλάμε για τον ενιαίο ουρανό, είναι περίεργο να μιλάμε για μπλοκ. Και από η διαδικασία που λέει να γίνονται διαγωνισμοί για υποψηφιότητες για ένα σχέδιο που αφορά τον ενιαίο ουρανό εμπεριέχει μια αντίφαση. Δηλαδή, από τη μια μεριά δημιουργείται εντύπωση ότι ας έχουν τα πράγματα και οι διαδικασίες σήμερα ακόμα δεν πάνε να μας οδηγήσουν προς ένα ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Και δεν είναι μόνο το εφέστη που δημιουργεί τα προβλήματα. Κύριε Πακένο, ερωτήσεις. 13 λεπτά περίπου σας μένουν για να ικανοποιήσετε την περιέργεια των συναδέλφων μου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους κύριους και κυρίες ευρωβουλευτές για τις ερωτήσεις που αντικατοπρίζουν και την περιέργεια της Επιτροπής σας και μια συζήτηση που γίνεται εδώ και μήνες, χρόνια για τη διαδικασία που θα μας οδηγήσει σε έναν ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Και τα λειτουργικά αυτά τμήματα φάμψη είναι ένα κομμάτι της διαδικασίας αυτής. Η εισαγωγή μου πριν και το σχέδιο απόφασης επιλογής που σας έχει υποβληθεί είναι μόνο ένα στοιχείο, μικρό στοιχείο του συνόλου αυτών των διαδικασιών είναι το πρόγραμμα RTT στο πώς θα βοηθήσει σιγά σιγά να υπάρξουν αυτά τα λειτουργικά τμήματα ενέργειου χώρου FABs. Είναι ένα κομμάτι μόνο μιας διαδικασίας και είναι μια διαδικασία bottom-up όπως τη λέμε στα αγγλικά. Δηλαδή το 2008 και το 2010 τώρα τα ενδιαφερόμενα κράτη, ενδιαφερόμενα για τα FABs, έκαναν προτάσεις Μερικές φορές ήταν απλώς ε, μελέτη σκοπιμότητας, σε άλλε περιπτώσει είχαμε μηχανισμούς διαβούλευσης και συντονισμού που διευκολύνονται από κοινοτική χρηματοδότηση και σε πολύ λίγε περιπτώσεις και επενδύσεις σε συστήματα και τεχνολογία που επιτρέπει να λειτουργούν αυτά τα λειτουργικά τμήματα του ενέργειου χώρου. Οι τέσσερις αποφάσεις χρηματοδότησης που είναι υπό μελέτη σήμερα δεν είναι η πολιτική του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού ούτε ένα αποκλειστικό στοιχείο στη δημιουργία αυτών των ΦΑΜ. Σας θυμίζω, ο στόχος είναι να ολοκληρωθούν αυτά μέχρι το τέλος του 2012 και η χρηματοδότηση RTET στοχεύει στο να διευκολύνει αυτό το εγχείρημα. Και έτσι απαντάω σε μερικές ερωτήσεις. Γιατί είπαμε χάρη, γιατί περισσότερα χρήματα για το Α και όχι για το Β γιατί ορισμένα FAB καλύπτονται και ορισμένα όχι. Αυτό αντικατοπτρίζει τις προτάσεις που μας υπέβαλαν τα κράτη-μέλη με βάση το πρόγραμμα εργασίας που ετοιμάσαμε στις αρχές του χρόνου. Το περιεχόμενο αυτών των προτάσεων ποικίλει. Μία πρόταση που υποστηρίζει το FAB FABEC έχει ποσό πολύ πιο μεγάλο από ό,τι άλλες προτάσεις. Φυσικά εμείς το 2008 χρηματοδοτήσαμε και οι αποφάσεις συνεχίστηκαν και για το 2009, αποφάσεις όμως το 2008 ήταν, πέντε FABs. Κεντρική Ευρώπη, 2 εκατομμύρια, Blue Med με Ιταλία, 2,8 εκατομμύρια και αυτό εξηγεί γιατί αυτοί που έκαναν τον απολογισμό έκαναν ότι η πρότασή μας δεν ήταν εντελώς όριμοι ένα πρόγραμμα North European ATM Concept 800.000 ευρώ Τι στα έχουμε μια μελέτη για το Δούναβι, το FAB 2,5 εκατομμύρια και τέλος μια μελέτη σκοπιμότητας για να γίνει ένα FAB της Βαλτικής 1 εκατομμύριο αυτό προτείνεται σήμερα μάλλον θα πρέπει να συγκρίνεται αυτό που προτείνεται σήμερα με τις αποφάσεις 2008-2009. Και όλα τα προγράμματα αυτά τρέχουν ακόμα σήμερα από ό,τι ξέρω. Θα αρχίσω με το ερώτημα του κυρίου Γκρός για τα κριτήρια. Υπάρχουν στο πρόγραμμα εργασίας, καλό να μπουν και στο μπροσούρα στο φυλάδιο είναι να relevance της πρότασης, να έχει νόημα η πρόταση και θα συνεχίσω στα αγγλικά γιατί έχω στα αγγλικά το κείμενο. Οι προτάσεις θα πρέπει να είναι εύστοχες και να πληρούν τις προδιαγραφές του FAB με σχέση με στόχο τον Ευρωπαϊκό Ουρανό. Πρέπει να υπάρχει απόδειξη ότι το πρόγραμμα μπορεί να μέχρι το 2012 να είναι εφαρμόσιμο. Αυτά τα προγράμματα που είναι αξιόπιστα με προθεσμία 2012 αυτά θα χρηματοδοτηθούν. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν και άλλα πράγματα. Θα επανέλθω σε αυτό. Η οριμότητα του προγράμματος, οι διάφορες δραστηριότητες που καλύπτουν από την πρόταση θα πρέπει να είναι δυνατόν να εφαρμοστούν άμεσα. Η επίπτωση, και εδώ έχουμε κριτήρια, που είναι τα κλασικά κριτήρια του ενιαίου ουρανού, ποσοστό αύξηση στην αποδοτική χρήση των πτήσεων, ε, άριστη χρήση του δυναμικού κλπ. κλπ. Μετά έχουμε τα συνήθη κριτήρια ποιότητας. Είναι πλήρης, η δομή του management είναι σαφής και πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα είναι δυνατόν να εκτελεστεί λειτουργικά με την υπάρχουσα υποδομή. Αυτά είναι μερικά από τα κριτήρια που υπήρχαν και στο πρόγραμμα, αλλά πολύ ευχαρίστως να σας τα δώσω το απόγευμα σε, σε ένα φύλλο χαρτιού, να το έχουν οι βουλευτές μπροστά τους, θα είναι χρήσιμο. Δεύτερη ερώτηση του κυρίου Γκρός. Ποιο είναι το περιεχόμενο αυτών των προτάσεων. Εμείς το φυλάδιό μας το κάναμε βάσει του τι έγινε το 2008 στο φυλάδι θα έπρεπε να έχουμε πολύ περισσότερες προτάσεις. Δεν είχαμε χρόνο να το κάνουμε για να μπούμε σε λεπτομέρειες. Πάντως είναι εύστοχο το σχόλιο του κυρίου Γκρός. Όχι μόνο να πούμε γιατί επιλέξαμε αυτά τα προγράμματα και πώς τα αξιολογήσαμε, το σημειώνω αυτό, ότι στοιχεία για το περιεχόμενο και την ουσία είναι χρήσιμα. Αυτό που μπορώ να σας δώσω το απόγευμα ήδη η εσωτερική αξιολόγηση, τα σχετικά φύλλα που υπάρχουν για κάθε πρόταση από τη μέση τρει-τέσσερι σελίδε για το καθένα, έχετε το περιεχόμενο, την συγκεκριμένη δραστηριότητα, τα κονδύλια που δόθηκαν και η αξιολόγηση και από τους εξωτερικούς συμπεριγνώμενους και από το πάνελ της Κομισιόν. Αυτό το κάναμε και στο παρελθόν. και θα σας δώσουμε τις έξι αυτές εκθέσεις με όλες τις λεπτομέρειες. Για τα κονδύλια για τα φάμψη ήδη απάντησα, σας τα είπα πριν τα νούμερα και αν θυμάμαι το 2008 δαπανίσαμε 20 εκατομμύρια. Λάθος, το 2008 10 εκατομμύρια. Τώρα έχουμε 20 διαθέσιμα για, για αυτές τις προσφορές τώρα. Υπάρχει μια αναλογία μεταξύ των ποσών που δίνονται και την δέσμευση, την δυνατότητα των κρατών μελών να υλοποιήσουν τα FAB μέχρι το 2012. Όχι, όχι, δεν υπάρχει τέτοια αντιστοίχηση. Η λογική του να δίνονται τα κονδύλια στηρίζεται μόνο στην πρόταση αν ζητάτε κονδύλια και οι δραστηριότητε συμφωνούν με τα κριτήρια, θα δοθούν τα χρήματα. Όταν κάνουμε μια αξιολόγηση εκ των υστέρων, ναι, εκεί κοιτάμε. Ήταν χρήσιμα, χρησιμοποιήθηκαν με σωστό τρόπο τα κονδύλια αυτά ή όχι. η προθεσμία του 2012 θα τηρηθεί, ερώτησε η κυρία Γιάνσεν. Το συζήτησα με τους συναδέλφους, ενώ θέτετε το ερώτημά σας και απαντώ. Οι ε, κατευθυντήρες γραμμές του Eurocontrol θα τις έχουμε το φθινόπωρο, πάνω κάτω. Η διαδικασία είναι bottom-up, σας είπα η εικόνα συνεχώς αλλάζει, οι πληροφορίες από τις προσφορές μας το δείχνουν αυτό. από την άλλη μεριά δεν έχουμε δείξει ότι δεν θα πετύχουν να τηρήσουν την προθεσμία τα FAB. Με βάση την εμπειρία μου απάντησα στο σημείο αυτό. Αν υπάρχουν επιπλέον ερωτήσεις η Κομισιόν ευχαρίστως θα απαντήσει γραπτά σε πιο λεπτομερείς ερωτήσεις. Και όπως ξέρετε, συμφωνήσαμε να υπάρξει ένας συντονιστής για τα FAB που με τις κατευθυντήρες γραμμές, το guidelines, την χρηματοδότηση αυτή εδώ και τη δέσμευσή μας θα διευκολύνει την υλοποίηση των προγραμμάτων μέχρι το τέλος του 2012. Γιατί η Σλοβακία δεν συμπεριλαμβάνεται. Η Σλοβακία παραμένει στη διαδικασία αυτή της τώρα. Το, αν, το γιατί αποφάσισε να μην επιμείνει στην συμμετοχή μέσα στη συγκεκριμένη αυτή απόφαση χρηματοδότησης δεν μπορώ να απαντήσω αυτή τη στιγμή, θα το ελέγξω. Παραμένει στο λειτουργικό σκέλος πάντως η Σλοβακία για τα στρατιωτικά δεν θα απαντήσω γιατί δεν ξέρω τι ρόλο παίζει η βιομηχανία. Τα προγράμματα αυτά τα κάνουν οι υπάρχοι υπηρεσιών. Άρα η βιομηχανία παίρνει μέρος. Αλλά στις προσφορές έχουμε συγχρηματοδότηση, αυτούς παρέχουν τις υπηρεσίες, κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν θα γίνει λειτουργικό το ΦΑΜ, φυσικά εκεί ο ρόλος της βιομηχανίας θα είναι κεφαλαιώδης. Γιατί όχι το BlueMed χρηματοδοτήθηκε το 2008 και τρέχει όπως σας είπα το πρόγραμμα αυτό ήδη. Η κυρία Γιαλά ρώτησε γιατί η μερικά ΦΑΜ δεν έκανε πρόταση για χρηματοδότηση και συγκεκριμένα η Ισπανία-Πορτογαλία. Η απάντησή μου είναι ειλικρινά δεν ξέρω πιθανώς θεώρησαν ότι δεν χρειάζονται αυτή τη χρηματοδότηση μέσω προσφορών. Μπορούν να το κάνουν, να προχωρήσουμε το ΦΑΜ χωρίς τη διαδικασία αυτή προσφορών. Ε, πάση αυτό είναι η κασία δική μου. Θα πρέπει να δούμε οι αρχές τι έχουν να πούν για τις χώρες αυτές που δεν ζήτησαν χρηματοδότηση. Αν δείτε όμως τη χρηματοδότηση του 2008 και τη σημερινή, υπάρχει ευρία κάλυψη μπορούμε να πούμε για το πρόγραμμα 101 και το ποσοστό χρηματοδότησης. Το ποσοστό χρηματοδότησης είναι το επιλέξιμο κόστος και αν ε, ε, ε, χρηματοδοτούμε μελέτες ή έργο. Αυτό εξηγεί τα διάφορα ποσοστά. Τι επιμερισμός υπάρχει σε έργο και σε μελέτες. Κάπου μειώσαμε το εύρος του προγράμματος και αυτό επηρέασε το ποσοστό. Στο 42% που βλέπετε κάπου είχαμε περισσότερες εργασίες από ότι αυτές που ε, μεταξύ αυτών που προτάθηκαν και αυτός, αυτών που τελικά επιλέχθηκαν για την ενοποίηση των λειτουργικών τμήματων και τον λευκό χώρο στα Βαλκάνια. Αυτό αντικατοπτρίζει πρώτον το ότι η Σερβία, Μοντενέγκρο, η πρώην δημοκρατία, η Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και το Κόσοβο δεν είναι επιλέξιμη για τις προσφορές και δεν συμμετέχουν στο λειτουργικό τμήμα. Μπορεί να γίνει στο μέλλον. Ακόμα δεν συμμετέχουν. Η Βοσνία, Ζεγοβίνη και η Κροατία συμμετέχουν. Αλλά δεν είναι επιλέξιμες για τις προσφορές. Το ίδιο ισχύει και για άλλες τρίτες χώρες που μπορούν να πάνε μέρος στο εγχείρημα αλλά η χρηματοδότηση για τις προσφορές θα είναι μόνο για τις 27 χώρες μέλη. Δεν θα σχολιάσω γιατί το Μαρόκο και η Τουρκία δεν είναι μέσα. Λειτουργικά συμφωνώ και εγώ ότι έχει νόημα να είναι μέσα. Αλλά ο ενιαίος ευρωπαϊκός ε, ουρανός συζητιέται στα πλαίσια της ε, διαπραγματεύσεων με την Τουρκία συζητιέται με το Μαρόκ για, σε σχέση με την αεροπορική συμφωνία. Αλλά όπως σας είπα δεν είναι μέλη αυτή τη στιγμή ακόμα της διαδικασίας. Δεν απάντησα στην κυρία Μάιστερ. Ποια είναι τα ασθενή σημεία και γιατί χρειαζόμαστε τα FAMS. Η διαδικασία του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού που στηρίζεται στην ανάλυση αυτή και δεν ξέρω αν υπάρχει μια ενδιάμεση μελέτη αξιολόγησης που θα ορίζει τα κύρια ασθενή σημεία στη διαδικασία αυτή και προεδρεωτήσετε πώς εφαρμόζεται η συνεργασία για τα FABs. Εφαρμόζεται μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών των κρατών μελών και ημών της Κομισιόν. Έχουμε το πρόγραμμα των προσφορών που συζητάμε σήμερα, έχουμε το συντονιστή του FAB, Έχουμε την γενική πολιτική και δράση και τη συνεργασία κομισιών κρατών μελών. Επαναλαμβάνω, έχω την αίσθηση ότι δεν απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις, αλλά για όσε μπορούσα, για να σας πληροφορήσω, το έκανα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε